Καλημέρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 11, αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων εναντί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο συνάδελφος ε, Κέλλη, ο εισηγητής δηλαδή δεν είναι παρόν και θα αντικατασταθεί από τον συνάδελφο Ιντσού. Βρήκα ένα χαρτί, ένα φίλο χαρτί που μου λέει αυτό. Α, χαίρομαι. Α, είναι εδώ ο κύριος Κέλλη. Σας δίνω αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χτες έπαιζα μπάλα. Επέζησα. Οπότε να είμαι εδώ. Ε- η προστασία αυτή για τα φυσικά πρόσωπα είναι ίσως η πιο σπουδαία πρόταση που έχει περάσει αυτή τη θητεία. Ξεκίνησε αυτή η υπόθεση από το 1995 αλλά βέβαια από το 1995 έχουν πολλά αλλάξει. Επομένω. Και επιβάλλεται τώρα να γίνει κάποιο είδου ενημέρωση και κάποιο είδου φρεσκάρισμα. Έχουμε όμω έναν κανονισμό και έχουμε και μια οδηγία όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. αφορά τα ποινικά δικήματα κλπ. Είναι, είναι σημαντικός ο και είναι σημαντικό το ότι υπάρχει κανονισμός γιατί πρόσφατα είχαμε πάρα πολλές λαθροχειρίες σε σχέση με αυτά τα προσωπικά δεδομένα κυρίως μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά έχουν γίνει και, και άλλα θέματα όσον αφορά ας πούμε τις διαδικτυακές πωλήσει. Άρα, αυτό τώρα που χρειάζεται είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου. Και η Επιτροπή μας βεβαίω καλείται τώρα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε εξέλιξη στο μέτωπο των, της τεχνολογίας, ε, αυτών και των, και των, του Επίση, Επίσης, τα σχετικά το προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και το άρθρο 8 του Χάρτη των Δικαιωμάτων. Επομένως, μας περιμένει ένα έργο πολύ σημαντικό. Δε, γενικός ε, στόχος είναι να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τα τέλη της ε, τρεχούσης θητείας. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχουν πάρα πολύ χρόνο, αλλά οι σκιώδεις και ο εισηγητής θεωρούν ότι θα τα καταφέρουν. Θα πρέπει επίσης να απλουστεύσουμε τον νομικό και τους κανόνες, να μειώσουμε την γραφειοκρατία και να υπάρχει επομένως ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα. Να βγουν καινούργιες εταιρείε, να βοηθήσουμε τις υπάρχουσες και έτσι να βελτιωθεί η γενικότερη κατάσταση. Θα έχουμε επομένω έτσι ένα τέτοιο καινούργιο πλαίσιο, εμπιστοσύνη, καινοτομία, δημιουργικότητα. Επομένως, θεωρούμε ότι έτσι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και το ότι θα πρέπει να υπάρχουν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού, ιδίω για τι ΜΜΕ. Αλλά επίση αυτό αφορά και γενικότερα τη βιομηχανία σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε κάποιες προτάσεις Ήδη έχουμε συναντήσει 52 φορές διάφορους εμπλεκομένους, οπότε βλέπετε τι ενδιαφέρον υπάρχει από τον κόσμο και συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις. Επίσης ε, έχουν γίνει και διάφορες ε, συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για θέματα τεχνικά με τους συγκεκριτές. Ε, και τώρα σε σχέση με το κείμενο καθε αυτό έχουμε κάποια θέματα όπου θα πρέπει η Ήτρε να διαρματίσει σημαντικό ρόλο πρώτα από το οριζόντιο ζήτημα των ΜΜΕ. Η Ήτρε είναι η αρμόδια επιτροπή για όλα αυτά τα θέματα στο Κοινοβούλιο. Και επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις ΜΜΕ ότι να μην υποστούν αρνητικές συνέπειες από τον ε, κανονισμό αυτό. Και βεβαίω ενδιαφέρονται για αυτή την προστασία οι ΜΜΕ όπως και ενδιαφέρονται για αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Άλλο οριζόντιο θέμα αφορά την κοινωνία πληροφορία και την πληροφορική μια που έχουμε εμείς ρητή αρμοδιότητα άρθρο 8 και 90 βλέπουμε σχετικά και επίσης η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που είναι θέμα πάλι δικό μας. Γενικά αυτή η δημοκρατική πολιτική βεβαίως και είναι αποκλειστική μας αρμοδίωση με το άρθρο 22 που αφορά την συμμόρφωση, το 28 αφορά την τεκμηρίωση, το 33 ε, την μελέτη των επιπτώσεων, κεφάλαιο 3, το μήμα 4, το δικαίωμα προς ε, υποβολή ενστάσεων και γενικότερα ρυθμίσεις του άρθρου του κεφαλαίου 4 ε, επίσημη και το τμήμα υπαριθμών 4 Όλα, όλα, όλα αυτά τα τμήματα του κειμένου είναι ζητήματα αρμοδιότητα δική μα. Ήδη η πρόεδρο μα έχει απευθυνθεί στην πρόεδρο τη ΛΥΜΠΕ, ούτω ώστε να γίνουν διαπραγματεύσει και έτσι να ολοκληρωθούν οι επαφές και επίσης έχουμε δεσμευθεί να δουλέψουμε όσο πιο σκληρά γίνεται. Υποσχόμαστε να συναντήσουμε όσο γίνεται περισσότερο από του και επομένως να έρθει η μέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί ένας άρτιος κανονισμός ο οποίος θα προστατεύει τα φυσικά πρόσωπα αλλά επίσης θα δίνει το περιθώριο στις ε, ΜΜΕ να εξελιχθούν να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα και θεωρούμε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, γιατί ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και ότι η διεκπαιρέωση θα προχωρήσει τυχαίως. Ταχεία. Τώρα, επίσης, θα συνεργαστούμε, θα ακολουθήσουμε την πιο αποτελεσματική διαδικασία και υποσχόμαστε όλα αυτά να τα κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να σας πω, κάτι το οποίο αφορά την ε, μελέτη των επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε και σε αυτό το μέτωπο να κάνει ό,τι μπορεί. Υπάρχουν όμως εδώ πέρα κάποια προβλήματα. Πρώτα-πρώτα εδώ αναφέρεται το κόστος σαν ε, μία μεταβλητή και κατόπιν αναφέρεται το διοικητικό βάρος θεωρούμε ότι θα είναι σημαντικό πρόβλημα το διοικητικό βάρος. Επίσης, αναφέρονται θα πρέπει να δούμε το ρόλο των επιχειρήσεων, τι προβλήματα θα βρουν, γιατί εδώ πέρα αναφέρονται επίσης ο αποκλεισμό του χρηματοοικονομικού τομέα. Γιατί όλα όσα έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία 4-5 χρόνια οδηγούν σε αυτά τα προβλήματα του χρηματοοικονομικού τομέα. Και άρα θα πρέπει εδώ να είναι κανείς πολύ προσεκτικός λένε για το τι παραβιάσεις ε, αναμένονται να γίνουν όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Υπάρχει και πρόβλεψη στον κανονισμό για τον υπεύθυνο προστασία δεδομένων, DPO στα αγγλικά. Οπότε, ε, εάν κάνουμε μια ταχεία διεκπαιρέωση, θα έχουμε την προστασία ακόμα νωρίτερα, οπότε σας προτείνω σήμερα να δώσουμε το πράσινο φως για να προχωρήσει αυτή η πρόταση. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους που τον ζήτησαν, θα ήθελα να σας ενημερώσω σε σχέση με το ζήτημα του άρθρου 50. Όπως γνωρίζετε, εμείς ζητήσαμε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να εφαρμόζεται το άρθρο 50. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μας απάντησε αρνητικά, προτείνοντάς μας να χρησιμοποιούμε το άρθρο 49. Ακόμη και με διευρυμένη ε, ερμηνεία, ωστόσο επιμένει στη χρήση του 49. Ενημερώσαμε σχετικά, όπως γίνεται συνήθως, στη διάσκεψη των Προέδρων. Στην τελευταία του συνεδρίαση, η διάσκεψη των Προέδρων μας έδωσε τη σημερινή ημερομηνία ως τελική ημερομηνία για να επιτυχούμε μια συμφωνία. Εγώ συζήτησα χθες ε, στη διάσκεψη των συντονιστών μας και σε αυτή τη συνεδρίαση συντονιστών ε, υπήρξε κατά κάποιο τρόπο ισοψηφία μεταξύ όσων επιμένουν ε, στη χρήση του άρθρου 50 που ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες νομικές βάσεις ενώ υπήρχαν άλλοι σε σχέση με αυτό το ερώτημα ε, που ισχυρίζονται ότι μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόταση της ΛΥΜΠΕ γνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των άρθρων παρότι είναι σαφής η ερμηνεία πάντα δημιουργείται κάποια αντίθεση μεταξύ των δύο δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια λύση σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να ε, επιλέξει τελικά η διάσκεψη των Προέδρων. Στην επόμενη λοιπόν διάσκεψη των Προέδρων θα βρεθεί η λύση. Σήμερα αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα αίτημα από εμάς, άρνηση από τη ΛΥΜΠΕ, μια θέση δική μας μοιρασμένη 50-50 μεταξύ των όσων επιθυμούν το άρθρο 50 και όσων όχι. Έτσι λοιπόν η διάσκεψη των Προεδρών θα χρειαστεί να λάβει τη σχετική απόφαση. Ας προχωρήσουμε. Εγγεγραμμένοι ομιλητές ε, είναι ο κύριος Άλμπρεκτ, ε, εισηγητής της ΛΥΜΠΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους ε, της ε, κυρίας Τικάου και θα σας παρουσιάσω τις ιδέες της. Η προστασία των δεδομένων είναι σημαντική όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για ε, τον βιομηχανικό τομέα, τον οικονομικό τομέα. Θα πρέπει να φροντίσουμε ο οικονομικός τομέας να ενεργεί σύμφωνα με το πακέτο προστασίας δεδομένων. Είναι σημαντικό το πακέτο αυτό, όχι μόνο εντός ε, του εδάφους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ε, θεμελιώδες δικαίωμα. Θα πρέπει να έχουμε ενιαίους κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον βέβαια οι προϋποθέσεις αυτές ε, είναι, ε, συνάδουν με το Σύνταγμα των κρατών μελών. Ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων κινητικότητας ιδιωτική ζωή και οικογενειακής ζωής της ε, των την εμπιστευτικότητα του ιδιωτικού βίου θα, η ε, κυρία Τικάου τονίζει ότι με την ε, αύξηση της χρήσης ε, των υπηρεσιών cloud, του υπολογιστικού νέφους δηλαδή, Υπάρχει πρόσβαση από εξυπηρετητές σε δεδομένα άλλων ανθρώπων. οι ελεγκτές ε, θα πρέπει να έχουν διαφανείς ε, πολιτικές όσον αφορά την πρόσβαση ε, στα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ας αρχίσουμε τις παρεμβάσεις. Ο πρώτος εγγεγραμμένος, ο μιλητής, είναι ο συνάδελφος Ένσου. Ζητώ συγγνώμη. Έδωσα το λόγο στον κύριο Άλμπρεκτ πρώτα Πρώτα είχα δώσει το λόγο στον κύριο Άλμπρεχτ και μιλήσατε εσεί. Ε, κύριε Άλμπρεχτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Άλμπρεχτ, τον ε, ε, ε εισηγητή της ε, ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο παρότι δεν είμαι μέλος ε, της Επιτροπής σας. Ε, ανέλαβα την ε, πρωτοβουλία να παρευρεθώ διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό ήδη από την αρχή να συνεργαστούμε όσο γίνεται πιο στενά. Με τον κύριο Κέλλη είχαμε ήδη αρκετές συναντήσεις εδώ και ένα-δύο μήνες. Έχουμε ξεκινήσει τις τεχνικές μας συναντήσεις με την Κομισιόν και είχαμε και συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Έχουμε συζητήσει λοιπόν την πρόταση αυτή. Ως προς το περιεχόμενο, ο κύριος Κέλλη είπε ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα απλά να καταστήσω σαφές ότι είναι σημαντικό για μένα να σας πω ότι ε, ε, η ΛΥΜΠΕ ως Επιτροπή Αρμόδια επί της ουσίας ενδιαφέρεται να ε, συνεργαστεί στενά με τη δική σας Επιτροπή και με άλλες επιτροπές που ενδεχομένως θα γνωμοδοτήσουν για την έκθεση αυτή και θέλουμε όσο γίνεται νωρίτερα να οργανώσουμε τις συναντήσεις μας ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν όσοι εργάζονται πάνω στις σχετικές γνωμοδοτήσεις. Στην ε, Επιτροπή Προέδρων των Επιτροπών θα ε, ληφθούν οι απαραίτητες ε, συζητήσεις. Και κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου θα συνεργαστούμε, ελπίζω, μαζί με τον κύριο Κέλλη και τους σκιώδεις εισηγητές της ΛΥΜΠΕ να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου ώστε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό πριν το τέλος ε, της θητείας μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το είπε και ο κύριος ε, Κέλλη. Αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται σύντομα. Εδώ και 17 χρόνια ε, υιοθετήθηκε η παλιά οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Υπάρχει ανάγκη για πιο ισχυρή εναρμόνιση τον κανόνα της προστασίας των δεδομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ιδιωτικό βίο. Ε, έχουμε ένα οριζόντιο πρόβλημα το οποίο θέλουμε να λύσουμε από κοινού και ε, προσβλέπω στην ε, καλή συνεργασία. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κόσκο. Ευχαριστώ, κύριε ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, υπάρχουν κάποιοι που θα ψηφίσουν όχι στην συμφωνία άκτα. Ε, ήθελα να πω ότι ε, επικροτώ μια ε, μεταρρύθμιση ε, των κανόνων προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω το αποτέλεσμα αυτό να γίνει όσο το γίνεται καλύτερο. Αλλά ο λόγος που ζήτησα το λόγο είναι ότι Έχω σημαντικές αντιρρήσεις σχετικά με την πρόταση αυτή και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Ε, και μάλιστα η αντίρρησή μου αφορά μια άλλη αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, την έρευνα. Πατρίδα μου είναι η Σουηδία. Και έχουμε πολύ καλή έρευνα στα φάρμακα. Έχουμε και σχετικό βιομηχανικό κλάδο. Ο λόγος που έχουμε τόσο υψηλή ποιότητα είναι ότι έχουμε πολύ καλές δυνατότητες ε, να κάνουμε έρευνας με βάση τα μητρώα που υπάρχουν. Ε, τα μητρώα της ε, Σουηδίας καλύπτουν εκατοντάδες χρόνια και περιέχουν πολλές πληροφορίες ε, κοινωνικού χαρακτήρα και που σχετίζονται και με την υγεία. Και έτσι λοιπόν είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς ε, την εξέλιξη σε επίπεδο ατόμου, καθότι έχουμε και ε, προσωπικό αριθμό μητρώου. Η έρευνα αυτή ρυθμίζεται αυστηρά, υπάρχει στενή συνεργασία ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτές τις ιατρικέ έρευνε που να βασίζονται στα μητρώα. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις έρευνε αυτές, θέλουμε και άλλα κράτη-μέλη που έχουν αυτή την προσέγγιση να μπορέσουν να συνεχίσουν να ε, διεξάγουν τις έρευνε αυτές. Και έτσι τίθενται κάποια ερωτήματα η έγκριση της χρήσης των προσωπικών δεδομένων ε, στην έρευνα πώς ε, θα λειτουργήσει όταν ε, εργαστούμε με βάση αυτή τη νέα πρόταση. Από τη μία λέει ότι πρέπει πάντα να έχει κανεί την έγκριση το τόμο. Από την άλλη, οι απαραίτητες έρευνες θα εξαιρούνται από την απέτηση αυτή αλλά μπορεί αυτό να ισχύσει ε, για τόσο ευρεία χρήση δεδομένων ε, ε, ένας, ο μεγάλος όγκος είναι αποφασιστικός για τις έρευνες στη Σουηδία. Επίσης, το δικαίωμα να ξεχνιέται κανείς, το να διαγράψει δηλαδή τα δεδομένα του αποφασιστικής σημασίας για τις ε, ιατρικές έρευνες στη Σουηδία σήμερα είναι ότι μπορούν να διατηρηθούν τα δεδομένα για πολύ ε, μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι έρευνες αυτές οι οποίες ε, ε βραβεύονται και με βραβείο Νόμπελ και που, από τις οποίες αποφελούνται άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει και ο κανόνας ε, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων ε, ε, ανάλογα με με τη χρήση που προβλεπόταν κατά τη συλλογή των δεδομένων. Αλλά αυτό δεν είναι κανόνας που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην περίπτωση αυτή, διότι πριν 300-400 χρόνια έχουν, μαζευτεί κάποια, έχουν συλλεχθεί κάποια από τα δεδομένα αυτά. Ε, επίσης αναφέρεται η ηθική εξέταση για τις ιατρικές έρευνες αλλά και εδώ υπάρχει ασάφεια. Η πρόταση στην οποία θα καταλήξουμε ε, θα επιτρέπει τις έρευνες αυτές. Δεν θέλω να καταλήξουμε σε... στην κατάσταση όπου βραχυπρόθεσμα να έχουμε δυνατότητα για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας ε, στην χώρα μου, ε, αλλά μακροπρόθεσμα να ε, γίνουν τόσο αυστηροί οι νόμοι, ώστε να μην μπορούμε να εξετάζουμε τις ε, μακροπρόθεσμες ε, ε, συνέπειες ε, περιβαλλοντικών ε, τοξικών υλών ή να μπορούμε να εξετάσουμε την υγεία των παιδιών σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην πρόταση αυτή για τη δική μου αντιπροσωπεία και γι' αυτό πήρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Νίμπλερ. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή μας ε, Σον Κέλλη για την παρουσίασή του. Ε, δυστυχώς πρόλαβα μόνο το τέλος της παρέμβαση του, διότι έφτασα λίγο αργά. Αλλά θα ήθελα καταρχήν να πω ότι βρίσκω την ιδέα μελέτης αντικτύπου εξαιρετική και θα ήθελα να συμφωνήσω με την ιδέα αυτή. Βρίσκω ελπίσεις ε, ε, εξαιρετικό το ότι παραβρίσκεται ο συνάδελφος Άλμπρεχτ. Ε, και άσχετα από το αν επιλέξουμε το άρθρο 49 ή 50 ως βάση για την συνεργασία μας, πιστεύω ότι είναι θετική η συνεργασία ανάμεσα στις Επίτροπες στην Επιτροπή μας. Είχαμε πολύ θετικές ε, εμπειρίες στην Επιτροπή μας από συνεργασία με, άλλα, με άλλες αντιπροσωπείες, όπως για παράδειγμα ε, ε, στο θέμα της περιαγωγής. Βρίσκω λοιπόν εξαιρετικό το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα και μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν να προχωρήσουμε στην πλήρη εναρμόνιση ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό στην Ευρώπη να έχουμε ενιαίους ε, κανόνες ε, στην Ευρώπη. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κανονισμό και όχι Θα ήθελα στον εισηγητή να πω ότι από γερμανικής πλευράς θα πρέπει να προσέξουμε φυσικά η πλήρης εναρμόνιση να συνάδει με το Σύνταγμά μας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια νομική γνωμοδότηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, αλλά ε, δικαστές ε, του, του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου έχουν πει ότι η πλήρης εναρμόνιση δεν συνάδει με το Γερμανικό Σύνταγμα. Θα ήθελα να αποφύγω να ε, έχουμε να υιοθετήσουμε εδώ έναν πολύ ωραίο κανονισμό, ο οποίος όμως ε, τελικά σε δεύτερο στάδιο ε, να μας δημιουργήσει προβλήματα στη Γερμανία. Παρακαλώ λοιπόν τον εισηγητή να εξετάσει μήπως μπορούμε να έχουμε νομική γνωμοδότηση ώστε να μην παραβιάσουμε το Σύνταγμα καμιάς χώρας. Αυτό άλλωστε ήταν, δεν θα ήταν επικοδομητικό. Επίσης ήθελα να πω ότι βρίσκω καλή την πρόταση αυτή. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στις αρμόδιες επιτροπές και θα πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, όμω, ε, να μην ε, ε, ε, πνίξουμε τις ε, μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις με ε, υπερβολικούς κανόνες, να μην έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να αναπτυχθούν στο διαδίκτυο οι επιχειρήσεις αυτές. Από τη μία δηλαδή θέλουμε υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, από την άλλη μεριά θέλουμε να επιτρέψουμε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας να αναπτυχθούν οικονομικά. Νομίζω ότι σε πολλά επιμέρους θέματα θα πρέπει να έχουμε σχετικές συζητήσεις στην Επιτροπή μας. Για παράδειγμα, ε, βρίσκω πολύ καλές ε, τις ε, συζητήσεις για το Privacy by Design καθώς και το Privacy by Default. αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μελέτη αντικτύπου του Κοινοβουλίου, όπως είπα, για να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη, ώστε να φροντίσουμε να μην δημιουργήσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα ήθελα πολύ να, ήταν, να είχαμε και πυρογνώμονες εδώ που θα μπορούσαν να μας μιλήσουν για το profiling. Το ερώτημα είναι τι επιτρέπεται, πού θα πρέπει να προσέξει κανείς για να, φροντίσει, για, για να αποφύγει να γίνεται τέριασμα των δεδομένων ε, Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ε, πληροφορίες, δηλαδή τι γίνεται στην πράξη και ε, τι έχει νόημα να ρυθμίσουμε εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τρίτη παρατήρηση, ε, δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί κάποια ακρόαση, αλλά στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι στόχος μας να παραμείνουν οι επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη και όχι με αυστηρούς κανόνες προστασίας δεδομένων να οδηγήσουμε τις επιχειρήσεις σε μετεγκατάσταση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν συλλέγονται στοιχεία στην Ευρώπη, Μάλλον θα πρέπει να αποφύγουμε τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στην Ευρώπη από μια επιχείρηση να χρησιμοποιούνται εκτό ε, τη Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνε εντό και εκτό Ευρώπη για τα δεδομένα που συλλέγονται εντό τη Ευρώπη. Ε, είναι πολύ σημαντικό ε, συλλογισμό τον οποίο ήθελα να παρουσιάσω. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις ε, επιχειρήσεις μας ε, στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο πακέτο στο τέλος. Προσβλέπω στην ε, καλή συζήτηση και είμαι πεπισμένη ότι το θέμα βρίσκεται σε, πολύ καλά χέρια στα χέρια του εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Sí, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι καλή η πρόταση της ε, Κομισιόν και επικροτώ την ε, συζήτηση για επικαιροποίηση των ε, κανόνων η Ευρώπη θα πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων και είναι σημαντικό ε, και για τους Ευρωπαίους ε, καταναλωτές ε, και για τους παρόχους υπηρεσιών, για παράδειγμα, στο ψηφιακό περιβάλλον. Είναι σημαντικό η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων να γίνεται με διαφανή τρόπο. Πιστεύω ότι υψηλά πρότυπα σε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων ε, κάλλιστα μπορεί να συμβάλλει σε ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Του, του λεχθέντος είναι επίσης σημαντικό ε, να προστατεύσουμε την ε, δυνατότητα ε, να γίνονται έρευνες με βάση τα μητρώα που υπάρχουν. Θα ήθελα να συμφωνήσω δηλαδή με την συνάδελφό μου Ουλσκογ. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τους τρόπους να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Προσβλέπω στη συζήτηση που μάλλον θα κρατήσει πολύ καιρό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι ομιλητές. Δίνουμε τον λόγο λοιπόν στον κύριο Βέρμπικ από την Επιτροπή. Παρακαλώ. Ähm, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επικροτούμε ε, τις ε, γνώμες ε, των βουλευτών. Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί τους. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν καλύπτει πολλές από τις στοιχές που ήδη αναφέρατε σήμερα. Όσον αφορά την εξισορρόπηση δηλαδή του ε, συμφερόντος του ατόμου, να έχει δηλαδή υψηλό επίπεδο ε, προστασίας των δεδομένων και από την άλλη σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, των, ανθρώπων και από την άλλη να φροντίσουμε να μην επιβάλλουμε ε, παράλογο διοικητικό άχθος στις ε, επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε την ισορροπία αυτή και υπάρχουν και διατάξεις στην πρότασή μας και για την έρευνα που γίνεται με βάση τα, μητρώα, τα υπάρχοντα μητρώα. Με λίγα λόγια, ε, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την συνεργασία, ε, τη συζήτησή σας και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Κέλλη, έχετε πάλι το λόγο. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ενδιαφέροντα είπαν. Τους ευχαριστώ και γενικά μπορώ να πούμε ότι όλοι έχουμε υποσχεθεί να καταλήξουμε σε κάποιο δίκαιο, ισορροπημένο αποτέλεσμα, προστασία του φυσικού προσώπου, αλλά επίσης να εξασφαλίσουμε και την ε, πρόοδο της επιχειρηματικότητας και βέβαια και ως ε, Ήτρε ε, έχουμε υποχρέωση προς την βιομηχανία να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Οπότε και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα διαβιβάσουμε στον ε, εσύ τον κύριο Άλμπρεχτ τι έγινε ε, για τον Σουηδοφίλο επίση θέλω να πω ότι είναι σημαντικά τόσα είπε για την ε, έρευνα στην ιατρική πώς θα γίνει να μην έχουμε φραγμούς σε αυτή την πορεία δεν θα πρέπει να θεσπίζουμε μονοθετήματα τα οποία εμποδίζουν. Ό, όσα είπα θα τα λάβουμε υπόψη. Και η κυρία Νίμπλερ είπε σημαντικά. Την ευχαριστούμε για την υποστήριξή της σε σχέση με τη μελέτη των επιπτώσεων. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα επιμείνουμε να θεσπιστεί τελικά κανονισμός και όχι η οδηγία που θα ήταν λάθος. Δεν θα βοηθούσε σε αυτό το στόχο που έχουμε. Βεβαίως και οι ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικές και ε, η Άγγελα ανέφερε το ότι ίσως χρειαστεί να κάνουμε ακροάσεις. Ναι, θα το έλεγα και εγώ αυτό. Ήδη το έχουν πει κάποιοι από τους ε, εμπλεκόμενους ή θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους εμπειρογνώμονες. Και τελικά γι' αυτό να έχουμε μια ισορροπημένη προβληματική. Επομένως, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις. Θέλουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα υψηλό επίπεδο αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Οπότε Γι' αυτό τελικά με Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εισηγητή θα υπάρξει συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλε γνώμε, να έχουμε έναν αξιόλογο κανονισμό και να αποφύγουμε τι ε, αρνητικέ ε, συνέπειε. Γιατί δεν θέλουμε τελικά αντί για καλό να κάνουμε κακό με αυτόν τον κανονισμό. Σα ευχαριστώ. Grazie. Ε, Ευχαριστούμε στην Κέλλη. Ακόμα δεν έχουμε τις ημερομηνίε για την ε, επόμενη συζήτηση του θέματος. θα δούμε τι θα γίνει με το σχέδιο γνωμοδότησης και κατόπιν θα κανονιστεί η ημερομηνία σχετική και θα σας ε, ενημερώσουμε σχετικώς τώρα. Με την ευκαιρία του, της ώρας που μας περισσεύει πριν την ψηφοφορία μπορώ να σας πω τι έγινε χθε το βράδυ στις συνεδρία των συντονιστών. Προγραμματίσαμε τις ε, συναντήσεις μας τον Σεπτέμβριο. Δεν θα γίνει η συνάντηση της 6 Σεπτεμβρίου γιατί υπάρχει μια επικάλυψη με τις ε, ημέρες, ημερίδες μελέτες του ΕΛΚ. Επομένως θα γίνει συνάντηση στις 3 Σεπτεμβρίου, 15 με 18 και στις 30 θα συζητήσουμε το σχέδιο νομοδότησης για τον προϋπολογισμό του... Στη συνέχεια στις 17 Σεπτεμβρίου το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 6.30 και 18 Σεπτεμβρίου όλη την ημέρα. Ουσιαστικά υπάρχει αυτή η αλλαγή του ημερολογίου ώστε να ε, καλύψουμε την ε, ημέρα της 6 Σεπτεμβρίου που δεν θα γίνει η Επιτροπή Ήτρε. Θα αφήσουμε την 7η Σεπτεμβρίου και θα έχουμε 3η, 17, 3 Σεπτεμβρίου 17 και 18. Όσον αφορά τις δημόσιες ακροάσεις, κατά το δεύτερο εξάμεινο του έτους μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου θα έχουμε μία παρουσίαση για τις βασικές τεχνολογίες και enabling technologies Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα γίνει το ίδιο για τα smart cities, της εξυπνες πολης πόλεις. 17-18 Σεπτεμβρίου για τον οδικό χάρτη για την ενέργεια για το 2050. Αντιθέτως θα αναβάλουμε για το 2013 την διαστημική πολιτική και για τα τέλη του έτους με συντονισμό της Επιτροπής ΦΕΜ το ε, θέμα για τις γυναίκες και το ICT. Παρακαλώ τον συνάδελφο Ρόιλ. Μία ερώτηση είχα. Έχω. Είπατε 18 Σεπτεμβρίου θα γίνει πρόσθετη ε, συνεδρίαση και είπατε ότι 17 και 18 θα γίνουν ακροάσεις. Δεν κατάλαβα. Και 17 και 18 θα έχουμε συνεδρίαση. Και τις δύο μέρες. Ευχαριστώ. Ε, Καταλάβατε σωστά. 17 και 18 Σεπτεμβρίου. 17 Σεπτεμβρίου. Μόνο το απόγευμα. 17 Σεπτεμβρίου από 3 το μεσημέρι έως 6 και μισή το απόγευμα. Και 18 Σεπτεμβρίου από 9 μέχρι 12.30 και από 3 μέχρι 6.30. Αυτές είναι οι νέες ημερομηνίε ε, στις οποίες προσθέθηκε η 3η Σεπτεμβρίου μόνο το απόγευμα από 3 μέχρι 6.30 και δεν έχουμε πλέον 6η Σεπτεμβρίου. Η 6η Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα μελέτης του ΕΛΚ. Δεν θα γίνει λοιπόν συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε. Θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, 17 το απόγευμα και 18 όλη την ημέρα. Άλλη πληροφορία ε, σε σχέση με τις συνεδρίες των συντονιστών. Η Επιτροπή ΣΤΟΑ πρότεινε να υποδείξουμε μέσω των συντονιστών τυχόν προτάσεις μελέτης έως την 5η Ιουνίου του 2012. Εάν θεωρούμε ότι πρέπει να υποδείξουμε μέσω των συντονιστών μας προτάσεις μελέτης, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι την 5η Ιουνίου. Ταυτόχρονα η ΣΤΟΑ κάλεσε για τις ε, ημέρες από την 11η έως 15η Ιουνίου στο Δουβλίνο υπάρχει ένα φόρουμ ε, στο οποίο θα, για το Euroscience στο οποίο θα συμμετέχουν οι συνάδελφοι Καρβάλιο και Τόμψον συγγνώμη 11 με 15 Ιουλίου όχι Ιουνίου δεν διερεμήθηκαν εκθέσεις κανένας είδους απλά αποφασίστηκε να αφήσουμε στο συνάδελφο Έρτσοκ τη συνέχιση των εργασιών για το δημοσιονομικό πλαίσιο με το οποίο ασχολείται ήδη. Αυτά είναι όλα όσα αποφασίστηκαν χθε στη συνεδρία των συντονιστών. Έχουμε τώρα 6 λεπτά διάλειμμα και στις 10 θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Bene, cominciamo Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Ε, έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Σας προσπαθήσουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε εγκαίρως, στην ώρα μας. Παρακαλώ καθίστε, βρείτε τις κάρτες σας. Ποιος θέλει μια ημέρα ηλιόλουστη στις Βρυξέλλες. Ψηφίστε όσοι θέλετε μια ηλιόλουστη μέρα στις Βρυξέλλες. Ψηφίστε. Εγκρίνεται. Λείπει ακόμα πολλοί κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Με την ε, ε, γνωμοδότηση Κράμερ.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 αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ε, άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Bene. Ωραία λοιπόν. 46 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερη, δεύτερος φάκελος ε, του εισηγητή κ. Κράμερ, τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρινέται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρινέται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4, 14 υπέρ, όχι 14, κάνει λάθος η πρόεδρος, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές Φαίνεται να απορρίπτεται. Ας το επαληθεύσουμε. Ε, Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 30. Κλείνει η ψηφοφορία. 29 υπέρ, 24 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά Αποχές. Φαίνεται να απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε. Για το 33, τροπολογία 33. Έχουμε δύο αριστερούς παραπάνω. Ε, μία, ε, ένα. 33, τροπολογία 33. 30 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 σε τρία μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές φαίνεται να εγκρίνεται ας κάνουμε έναν έλεγχο για την τροπολογία 10 Κλείνει η ψηφοφορία. 37 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 42 σε, 3, σε 4 μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 περ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία Κλείνει η ψηφοφορία. 50 υπέρ, ένας κατά, δύο αποχές, εγκρίνεται. Ο κύριος Μπιουτικόφερ. Συγχαρητήρια στον ε, εισηγητή. Έχουμε τώρα τη γνωμοδότηση Μπουτικόφερ για τον προπολογισμό. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία. Ζητώ συγγνώμη. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος της τροπολογίας 8. Τροπολογία 9. Δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 14 ε, συγγνώμη σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 σε δύο μέρη πρώτο τροπολογία 18 μόνο το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 23 υπέρ κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά απο, αποχές φαίνεται να εγκρίνεται ας το ελέγξουμε την τροπολογία 25 Χιούζα. Πέρας ψηφοφορίας 43 43-114 14 εγκρίνεται Συμβιβαστική 4 υπέρ. Παρακαλώ, συναδελφέ Μπιούτικοφ. To... Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να προτείνω μια προφορική τροπολογία, ούτω να αλλάξουν κάπως τη διατύπωση για αυτή τη συμβαστική. Αντί το κείμενο το οποίο λέει Ευρωπαϊκή Πράσινη Οικονομία, να ψηφίσουν το κείμενο που θα λέει η φορεία βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και αυτό έχει ζητηθεί από και συμφωνηθεί από τις πολιτικές ομάδες. Σύμφωνουν με όλοι να δεχθούμε την προφορική τροπολογία. Ωραία. Ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 4 με την, τροπολογία, την προφορική υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά αποχές Ελέγχουμε. Κλείνει η ψηφοφορία. 29 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 50 υπέρ. Επτά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια. Περνάμε στη γνώμη... Περνάμε στην ε, γνωμοδότηση. Συμβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ, 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική υπέρ κατά τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ ε, ε, λείπει 72 τροπολογία βρισκόμαστε στην έκθεση Τικάου 72 τροπολογία λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ τροπολογία 20 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές φαίνεται να απορρίπτεται ας το ελέγξουμε για την τροπολογία 25 της έκθεσης για το πρόγραμμα Creative Europe κλείνει η ψηφοφορία 31 υπέρ 26 κατά εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κα, κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ 29 συγγνώμη όχι 9 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστη... τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 54 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση συγχαρητήρια. Έχουμε την γνωμοδότηση Anders Dotter. Έτσι βάζουμε μαζί τις ψηφοφορίες τροπολογία 1, 2 και 14. Ψηφίζουμε μαζί για αυτές τις τρεις τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, απορρίπτονται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Έλεγχος για τροπολογίες 1, 2 και 14. Μαζί. έχουμε έναν σοσιαλιστή παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Έναν σοσιαλδημοκράτη παραπάνω. Ακόμη περισσεύει ένας. Υπάρχει ένας παραπάνω. Ωραία λοιπόν. Τέλεια αποτέλεσμα. 26 υπέρ, 31 κατά και απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μαζί. Τροπολογίες 3, και 4 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται ελέγχουμε ηλεκτρονικά για μένα είναι το ίδιο με πριν μικρή διαφορά υπάρχει αλλά στο ελέγξουμε ένα σοσιαλδημοκράτης παραπάνω υπάρχει ωραία αποτέλεσμα 26 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται και η τροπολογία 3 και 4. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Ας ψηφίσουμε για την τροπολογία 7 γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω ποιος είναι υπέρ ποιος είναι κατά. Τροπολογία 7 ψηφίζουμε τώρα. Κλείνει η ψηφοφορία. 18 υπέρ, 0 κατά, 38 αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ελέγχουμε την 23 ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. 33 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, α, ελέγχουμε την 6. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 6. Κλείνει η ψηφοφορία. 33 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 26. Κλείνει ψηφοφορία. 32 υπέρ, 23 κατά. Συμβιβαστική 3 απορρίφθηκε. Συνεπώς πρέπει να ψηφίσουμε και για τις επιμέρους τροπολογίες. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Ζητώ συγγνώμη, η συμβιβαστική 3 απορρίφθηκε. Έτσι λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε τις επιμέρους τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη, θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Παράγραφος 6. Υπέρ κατά Αυτή η τροπολογία δεν έχει αριθμό, είναι μόνο η παράγραφος 6, draft opinion. Ωραία λοιπόν, υπέρ, ε, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. «29 υπέρ, 26 κατά, άγκρινεται» appunto noi. Dopo tante prove. Sorry, Chair. Can you repeat the result, please? Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να επαναλάβετε το αποτέλεσμα. Περνάμε πάλι στο σχέδιο γνωμοδότησης, λέει η, η Πρόεδρος, συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ακόμη μια ψηφοφορία πριν από την τελική ψηφοφορία εκεί όπου γράφει recommendation, σύσταση όπως προηγουμένως και για το draft opinion Anders λοιπόν χωρίς αριθμό το βρήκατε ωραία θέτουμε σε ψηφοφορία αυτό υπέρ κατά αποχές δεν γνωρίζουμε Κανείς από τους δυο μας ε, το ελέγχουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Κλείνει η ψηφοφορία. 29 υπέρ, 25 κατά, 2 αποχές, έγκρινεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την γνωμοδότηση της Αμέλη Άντρες Ντότερ. Una notizia c'è una nomina di un municipalità. infatti che avevo un po' la testa via, per quello sono riuscita a telefonare. Franco. Bene, voto chiuso. Κλείνει η ψηφοφορία. Έχουμε ένα S&D παραπάνω. Έναν σοσιαλδημοκράτη παραπάνω από ό,τι πρέπει. Κλείνει η ψηφοφορία. 31 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. Allora, Franco. Φράνκο. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 και 35 μαζί υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 31 και 1 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ κατά, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι απορρίπτεται απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά Αποχές ε, μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Ας ε, ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 34. Κλείνει η ψηφοφορία. 32 υπέρ. 24 κατά. Εγκρίνεται τροπολογία. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 και 5 τροπολογίες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογίες 38 και 26 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογίες τροπολογία 16 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά. Τροπολογία 17 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά. Αποχές μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 18. Ελέγχουμε την τροπολογία 18. Votazione chiusa. Κλείνει η ψηφοφορία. 32 έναντι 20. Εγκρίνεται 42 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20-21 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 24, 4, συγγνώμη, 24, υπέρ. Κατά αποχές... Λοιπόν, εγκρίθηκε η 23, συνεπώς 24, 25, 23. έκανε λάθος ο πρόεδρος. Η 3 εγκρίθηκε, 24, 25, 23 καταπίπτουν, συνεπώς περνάμε στην 4 τροπολογία, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 53 υπέρ, ένα κατά, ε, εγκρίνεται συγχαρητήρια. Περνάμε στη γνωμοδότηση Σιμάνσκι. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ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 ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο να σας ε, επισημάνω ένα λάθος. Το λάθος που έγινε το εξή Το κείμενο της προφορικής τροπολογίας Δηλαδή έχουμε πρώτα η αρχική υπάρχει 15. Είπαμε, ο, ε, είπαμε θέλουμε να βγάλουμε μόνο την τελευταία φράση που λέει μεταξύ 80 και 95% από τώρα μέχρι το 2050. Το υπόλοιπο μένει ως έχει. Είναι όλα τα ίδια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι του κειμένου που ακυρώσαμε εμείς στην ψηφοφορία ουσιαστικά μένει. Απλά έχει διαγραφεί μόνο το τελευταίο μέρος 80-95%. Συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 15 με την προφορική τροπολογία έτσι όπως διευκρινίστηκε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1, 21 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ah, <coughs> Κλείνει η ψηφοφορία. 41 υπέρ, 1 κατά, 6 αποχές, συγχαρητήρια. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Ήμασταν πολύ γρήγοροι. Τα καταφέραμε πολύ καλά. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Αφήνουμε δύο λεπτά για όσους θέλουν να φύγουν από την αίθουσα ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε. Se possiamo riprendere i nostri Αν θέλετε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και παρακαλώ αυτοί που φεύγουν ας ε, βγουν με ησυχία. Σας παρακαλώ, λίγη στα γαλλικά η πρόεδρος. Μπορείτε να βγείτε. Και επομένως πάμε στο σημείο 23 της ημερησίας διατάξεως το 23. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή, τον κύριο Γκιούρκ, για να μας κάνει την εισήγηση της εκθεσεώς του. Έχετε το λόγο. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, tisztelt eh, kollégák, nem hiszem. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Τι, ό,τι να σας πω είναι λίγο όσον αφορά τη σημασία αυτού του θέματο. Ξέρετε πόσο σημαντικέ είναι αυτές οι δημόσιες συμβάσει. Όλοι το γνωρίζουμε. Πρέπει τώρα να σας ε, αναφέρω πάντω ε, κάποια στοιχεία ούτω ώστε να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η οδηγία. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε 50 ε, φορούς, φορείς που ασχολούνται με αυτές τις, ε, τις δημόσιες συμβάσεις πρώτη για το 18% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Έχουμε μόνος 2 εκατομμύρια ε, τέτοιες διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν συνολικά χώρα, επομένω βλέπετε ε, πόσο σημαντική είναι αυτή η οδηγία. Και ξεκίνησε αυτή η υπόθεση το 1971 και έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες ε, τροποποίησης, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν αλλάζουν. Ότι δηλαδή υπάρχουν κάποιες οριακές τιμές που τίθενται από αυτή την οδηγία και κατά τα λοιπά ισχύουν οι ποινικές διατάξεις. Τώρα η Επιτροπή έχει διπλό στόχο με αυτό το νομοθέτημα πρώτα-πρώτα να υπάρξουν κάποιες ε, ρυθμίσεις για να υπάρχει ε, υγιής ε, ανταγωνισμός. Και έχουμε τρεις αλλαγές που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος ζωής όταν γίνεται ο υπολογισμός και αξιολόγηση των προσφορών. Συμφωνώ. Διότι η τιμή αγοράς θα πρέπει να συνδυάζεται με την τιμή συντήρησης η οποία μπορεί να είναι ψηλότερη. Άρα, σε αυτή τη βάση θα γίνεται η αγορά. Δεύτερο. Το είδος της ε, διεξαγωμένης διαδικασίας. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξυγχρονιστεί η σημερινή διαδικασία και θέλει επομένω να επιφέρει κάποιες αλλαγές και να ισχύει μια νέα διαδικασία. Ε, τρίτο σημείο, τρίτος στόχος που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΜΕ. Σχετικά με τις ΜΜΕ θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει μια πιο ευέλικτη συμμετοχή. Και επίσης να έχουμε απευθείας πληρωμή στους υπεργολάβους. Αυτά όσον αφορά τις προτάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για τη δική μου ε, έκθεση να σας πω πώς δούλεψα. Επικέντρωσα την προσοχή μου σε διάφορα σημεία. Όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση στην ΙΜΚΟ την επίσης αρμόδια επιτροπή θα διαπιστώσουν ότι έλαβε υπόψη αυτό το οποίο και συζητήσαμε. Πάντω ε, πάντως στην έκθεση της ΣΥΜΚΟ δεν τονίζονται αυτά τα σημαντικά ζητήματα όσο θα έπρεπε. Πρώτα πρώτα. μη ε. Δεύτερον. Πράσινες αγορές και τρίτον η ανάπτυξη μιας ε, νέας κουλτούρας για τις, ε, για τις δημόσιες αυτές συμβάσεις. Όπως προείπα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μια πιο ευέλικτη ε, διαδικασία. Όμως δεν έχει διατυπώσει μια συγκεκριμένη πρόταση που να βοηθά στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φτάνει μέχρι το να προτείνει κάτι όσον αφορά τις δαπάνες, το κόστος το οποίο συνδέεται με τις, με τις δημόσιες συμβάσεις. Με πολλές φορές η συμμετοχή μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ. Ή τέλο πάντων τόσο να κοστίσει η τελο δημόσια σύμβαση. δημοσια όσον αφορά μια μικρομεσαία επιχείρηση, ε, αυτό το υψηλό κόστο μπορεί να τη ε, αποτρέψει από το να συμμετάσχει σε μια τέτοια δημόσια σύμβαση. Θα πρέπει να εξεταστεί ότι ισχύει σε κάθε κράτο μέλο. Και έχουμε εδώ πέρα ένα κατάλογο σε σχέση με το κόστος σε κάθε κράτος μέλος. Κάτι άλλο που επίσης αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ηλεκτρονική διαγωνισμία. Έτσι, οι έψιλων θα διευκολυνθούν αφού θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσει τους ηλεκτρονικά. Άρα θα έχουμε εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και επίσης θα έχουμε και λιγότερα λάθη. Έτσι επίσης θα υπάρχει διαφάνεια και καλύτερος έλεγχος. Αυτά όλα βρίσκονται στο κείμενο προ την Επιτροπή. Δεν θα έχουμε επικαλύψει, δεν θα έχουμε επανάληψη υποβολής των ίδιων ε, εντύπων. Όσον αφορά τις ε, πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τις ε, πράσινες αγορές, Είπαμε ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα βοηθήσουν να περάσουμε στην πράσινη οικονομία και θα είναι κάτι το οποίο θα καλύψει τις σχετικές ανάγκες της κοινωνίας μας. Δεν έχει προτείνει ούτε εδώ κάτι συγκεκριμένο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξάγονται τώρα διαπραγματεύσεις σε σχέση με την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Και εκεί αναφέρονται οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Και οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ αυτών των δύο νομοθετημάτων. Στην έκθεσή μας θέλουμε να υπάρχει συγκεκριμένη μνήμα πρώτα-πρώτα του ότι θα πρέπει όταν γίνεται η αξιολόγηση να την υπόψη το επίπεδο του κόστου ζωής και επίσης θα πρέπει να διευκολύνονται κάθε φορά να προτιμώνται όσα προϊόντα δεν οδηγούν σε υπερβολική κατανάλωση ενεργείας. Και η ΜΚΟ θα πρέπει να συντονιστεί βέβαια στο κείμενο της μαζί μας. Κάτι άλλο τώρα. Είπαμε πώς θα καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα καινούρια για τη σύμβαση δημοσίων συμβάσεων και εδώ στα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνώ. Έχω τι παρατηρήσεις παρατηρήσει σε αυτό το σημείο. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να υπάρχει μια κεντρική αρχή. Νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία, αν έχουμε ένα καινούργιο θεσμικό όργανο. Να συνεχίσουμε να έχουμε το σημερινό σύστημα, απλώς να το εφαρμόζουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έλεγχος εκτέλεσης. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει την προκήρυξη του διαγωνισμού, την πρόσκληση υποβολής ε, ενδιαφέροντος. Αλλά αφού μιλούμε εδώ για δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να τηρούνται εκτός από τις προθεσμίες και το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που προβλέπεται. Άρα θα πρέπει να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος στην εκτέλεση. Τρίτη παρατήρηση. Να άρουμε κάποια εμπόδια τα οποία υπάρχουν και εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των δημοσίων συμβάσεων. να υπάρξει προσαρμογή στην πραγματικότητα τη σημερινή και επίσης θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να διέπονται από αυστηροί, αυστηρούς κανόνες. Σήμερα έχουμε ένα σωρό περιορισμούς Οι τόσοι περιορισμοί οδηγούν σε παραδίαση των κανόνων. Ευχαριστώ να δεχθώ να λάβω υπόψη τις ε, προτάσεις και τροποποίησεις σας. Εγώ προσπάθησα να δώσω βάρος ε, σε αυτό που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας, ε, την πράσινη οικονομία, τις ΜΜΕ, και πάντως ε, ακόμα και για άλλο θέμα, αν έχετε μια τροποποίηση και άλλη τροπολογία, θα τροποποιήσω το κειμένο, ευχαριστώ να το λάβει υπόψη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να ακούσουμε τώρα τους σκιώδες ε, εισηγητές. Συνάδελφε Παλτσίδης, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας για τα πλήρη έγγραφά του και την παρουσίασή του. Δεν θα μακρηγορήσω πάνω στο θέμα αυτό, διότι θα μιλήσω ε, στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης ε, που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα. Όσον αφορά το έγγραφο αυτό, βλέπω θετικά την πρόταση της Επιτροπής ε, και τις προσπάθειες εξέβρισης σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην απλοποίηση των κανόνων και, ε, και των πολύπλοκων ε, διαδικασιών. Συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή όσον αφορά την ανάγκη των πράσινων συμβάσεων και θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην τιμή και την ποιότητα. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τις ε, συμβάσεις ως αποτελεσματικό εργαλείο της αγοράς. Μόνο όταν ε, όλες οι συμβάσεις ε, σε όλα τα κράτη-μέλη γίνονται ηλεκτρονικά, τότε θα μπορέσουμε να ε, πετύχουμε τον στόχο μας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ε, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες ε, δεξιότητες για την υποβολή συμβάσεων ηλεκτρονικά. Να σας πω ότι θα ήθελε η δική μου ομάδα να δει στην οδηγία. Θα θέλαμε μεγαλύτερη συμπερίληψη των κοινωνικών ε, πτυχών ε, όταν μιλάμε για ε, ανάθεση των συμβάσεων. τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια. Θα πρέπει να πληρούν και άλλα πρότυπα από τις συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, όσον αφορά τα κριτήρια για την απόρριψη προσφορών, θα πρέπει να γίνεται αυτό όταν η επιχείρηση παραβιάζει ε, κοινωνικά δικαιώματα ή πρότυπα ε, στην ε, αγορά απασχόλησης. Και τελευταία μου παρατήρηση, την οποία απευθύνω απευθείας προς την Επιτροπή, Όταν ε, μιλάμε για ανοιχτή αγορά δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να είμαστε τολμηροί και να προστατεύσουμε την αγορά μας από τρίτες χώρες οι οποίες ε, δεν ε, παρέχουν σε εμάς τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στη δική τους αγορά. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή την αρχή της αμοιβαιότητας ώστε ε, να μην ε, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι δικές μας επιχειρήσεις στις δικές μας αγορές. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Το λόγο έχει η κυρία Μάση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Μας δίνει μια αξιολογή αφετηρία για να προχωρήσουμε. Συμφωνώ με τη βασική του προσέγγιση, δηλαδή το να χρησιμοποιήσουμε τις ε, δημόσιες συμβάσεις ούτως ώστε να προχωρήσουμε προς μια συμμετοχική ε, και αηφόρο ανάπτυξη και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση της ενέργειας. Επίσης, συμφωνώ με την ε, προσέγγιση του να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το να χρησιμοποιείτε ε, το δημόσιο χρήμα με τρόπο ώστε να βοηθά την επίτευξη των ε, στόχων που έχουμε τάξει. Πάρα πολύ πάντως οι οποίοι ασχολούνται με την δύσμο συμβάσεις δεν καταλαβαίνουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτό το θεσμό. Τώρα ένα άλλο παράδειγμα ε, σημαντικό, το τι μπορούμε να πετύχουμε με τις ε, δημόσιες συμβάσεις είναι κάτι το οποίο συνέβαινε στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες επί Κλίντον. Αποφάσισε η κυβέρνηση ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αγοράζει υπολογιστέ μόνο εάν αυτοί ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας. Και αυτό επομένως ανάγκασε όλο τον κλάδο της κατασκευής υπολογιστών να γίνουν πιο αποτελεσματικοί ενεργειακά. Να, ένα καλό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει που είναι οι δημόσιες συμβάσεις, μια που είναι τόσο μεγάλος σημαντικός πελάτης στο κράτος. Τώρα, κάτι άλλο σε σχέση με αυτή την έκθεση, ε, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σχέδιο κειμένου σε σχέση με την ε, ενδιακή αποτελεσματικότητα. Σε αυτό θα πρέπει να γίνει πιο δυναμικό το κείμενο. Και ένας λόγος για τον οποίο θέτω το ζήτημα είναι το ότι είχα συμμετάσχει στις διαδικασίες σε σχέση με το αστεράκι, την ετικετοθεσία, τη σχετική με αποτελεσματικότητα και, και, και, και την ετικέτα της Ένωσης. Ε, θέλαμε ως Κοινοβούλιο να υποχρεούνται οι κρατικές αρχές να αγοράσουν ό,τι είναι πιο αποτελεσματικό ενεργειακά, ό,τι είχε το σχετικό αστέρι, ό,τι είχε τη σχετική ετικέτα για τον εξοπλισμό. Ό,τι, ό,τι τέλος πάντων ε, ήταν αγοραστή να, να, να, σχετίζεται να έχει αυτές τις ετικέτες. Και ε, το Συμβούλιο έλεγε ότι δεν είναι αντίθετη σε αυτό που λέμε, αλλά δεν είναι το σωστό μέρος να ρυθμίζεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει αυτό να προβλέπεται στην αντίστοιχη νομοθεσία για τη δημοσυμβάση. Ένα λοιπόν που τώρα έχουμε <clears throat> τη σχετική οδηγία. Επομένω, ο δωρητό μπορούμε να κάνουμε αυτή την πρόβλεψη. Όταν αγοράζονται κάποιε συσκευέ, να επιλέγονται πιο αποτελεσματικέ ενεργειακά. Κάτι άλλο τώρα. Ακόμα δεν είμαι βέβαιη, αλλά ε, σας ερωτώ, δεν ξέρω αν θα ε, ήταν σωστό να μην μονεύεται κάπως ε, σαφέστερα η αποτελεσματικότητα η ενεργειακή σαν ένα από τα κριτήρια για την ανοικοδόμηση κτηρίων γιατί άκουσα ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα από τις κάτω χώρες όπου τουλάχιστον ε, η πόλη του Άμστερνταμ για κάποια τέτοια έργα ε, καθόρισε την τιμή και ε, όταν έκανε τη δημόσια σύμβαση οι εταιρείε που ήθελαν να συμμετάσχουν θα έπρεπε να αποδείξουν πόσο αποτελεσματικό ενεργειακά θα είναι το κτίριο που θα φτιάξουν. Άρα μπορούμε και κάτι τέτοιο να βάλουμε στο κείμενο. Από ό,τι την έχουμε κάποιες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια προσώπων που αποφασίζουν ε, στον κρατικό τομέα για αυτές τις, ε, για αυτές τις, τις, τους διαγωνισμούς και αυτοί θα κληθούν μόνος να ε, ερμηνεύσουν το κείμενο. Ε, αυτοί ίσως μια φορά ε, βαριούνται να το ψάξουν βόλια και τελικά μπορεί να θεωρήσουν ότι έτσι τους πρόχουμε στο, στο, να αγοράσουν το πιο φτηνό. Δεν, δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει, ούτε εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά πολλές φορές ο κόσμος έτσι ερμηνεύει τα πράγματα. Τώρα το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να σας αναφέρω είναι αυτό το θέμα της, του ελαχίστου κόστους. Και ε, αντί, έχουμε τώρα αυτή την, την αρχή του ελαχίστου κόστου σε σχέση με την παλαιά αρχή της ε, κατωτάτης τιμής. Νομίζω ότι ε, θα οδηγηθούμε πάλι στο να ε, να, να έχουμε τον κανόνα του, της χαμηλότερης τιμής. Άρα θα πρέπει να αλλάξει εδώ η διατύπωση για να είναι σαφέστερη η νομοθεσία. Δηλαδή να είναι σαφές ότι το κόστος δεν είναι μόνο η τιμή αγοράς, αλλά και η τιμή, το κόστος της χρήσης. Τι γίνεται αφού ό,τι αγοράζεται, μηχάνημα, κτίριο, ό,τι να είναι, τι γίνεται με αυτό αργότερα ή όταν έχει κάνει τον κύκλο του, της, της χρησιμοποίησης του αυτό ε, το, ό,τι έχει αγοραστεί. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο πάλι ε, πάμε προς περισσότερη ποσότερο αποτελεσματική χρήση ενέργειας. Ευχαριστούμε τη συναρφάση. Το λόγο έχει ο συναδέλφος Ρόντερ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε αυτό που συζητάμε τώρα είναι να πραγματοποιήσουμε το e-procurement, τι ηλεκτρονικές ε, δημόσιες συμβάσεις, ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε την ενιαία αγορά. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για μια λειτουργική ενιαία αγορά. Οι δημόσιες συμβάσεις δηλαδή να πραγματοποιούνται ψηφιακά. Νομίζω επίσης ότι είναι πολύ λογικό να γίνει ε, υποχρεωτική εξέταση του κόστους κύκλου ζωής, ε, διότι μπορεί με την πρώτη ματιά να ε, είναι πιο φθηνό να βάλει κανείς μονό τζάμι στο παράθυρο, αλλά μπορεί αν εξετάσει κανείς τον κύκλο ζωής να διαπιστώσει ότι είναι πιο οικονομικό να χτίσει κανείς ένα κτίριο το οποίο να μην χρειάζεται ανακαίνιση μετά από λίγα χρόνια. Να εξετάσουμε δηλαδή ε, τις ε, δαπάνες που συνδέονται με το κύκλο ζωής. Ε, όσον αφορά τις ε, οριακές τιμές, τα κατόφλια, ε, υπάρχουν διστάμενες απόψεις. στη Δανία έχουμε διαπιστώσει ότι χωρίς να βλάψουμε την ενιαία αγορά, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το κατόφλι. Έχουμε το βασικό πρόβλημα ότι οι δημόσιες αρχές μας ε, ε, δαπανούν πολύ δυναμικό σε ε, διεθνείς διαγωνισμούς χωρίς να λαμβάνουν από άλλες χώρες προσφορές. Αυτό είναι σπατάλι δυναμικού. Μήπως λοιπόν να εξετάσουμε λίγο την πραγματικότητα και να συζητήσουμε τα κατόφλια. Διότι εμένα θα μου άρεσε να έχουμε κατόφλι στις ε, διεθνείς ε, συμβάσεις ύψους ενός εκατομμυρίου ε, ευρώ, διότι έτσι αξίζει τον κόπο να υποβάλει κανείς προσφορές από άλλες χώρες. Πολλές δημόσιες, πολλοί δημόσιοι διαγωνισμοί καταλήγουν στην κατάσταση όπου δεν λαμβάνουν προσφορές από το εξωτερικό και έτσι απλά έχουν σπαταλήσει πολύ κόπο. Όσον αφορά τις το δυναμικό του ε, δημοσίου τομέα. Ε, στόχος είναι η απλοποίηση της ε, διαδικασίας. Σε αυτό συμφωνούν όλοι, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε εδώ, διότι θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια απλοποίηση που να είναι τόσο δύσκολη η διαδικασία για αυτούς που υποβάλλουν τις προσφορές που τελικά να καταλήξουμε σε μια μη επικοδομητική λύση. Εάν κοιτάξουμε την πρόταση της Κομισιόν, Πιστεύω ότι η απλοποίηση γίνεται με λάθος τρόπο, διότι ουσιαστικά ανοίγει την πύλη ώστε οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιες αρχές μόνες τους να επιλέγουν σε ποιον θέλουν να αναθέσουν το, τη σύμβαση. Αυτό το πρόβλημα ήδη υπάρχει σήμερα. Αλλά Ε, θα πρέπει να δούμε με τα μάτια των επιχειρήσεων την ε, απλοποίηση που προβλέπετε. Όσον αφορά την ευθύνη και τα κοινωνικά κριτήρια που θέλουμε να εισάγουμε, εγώ είμαι επιφυλακτικός. Νομίζω ότι η ευθύνη για όλη την αλυσίδα παραγωγής ε, είναι πολύ κακή ιδέα. Δεν, θεωρώ ότι μπορεί κανείς να κάνει υπεύθυνη την εταιρεία για τις πράξεις όλων των ε, υπεργολάβων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα όλων των άλλων επιχειρήσεων, κάτι που θα καταστήσει αδύνατη την ε, διατήρηση ε, μυστικών των επιχειρήσεων. Και αυτό ισχύει και για τα κοινωνικά κριτήρια. Ανοίγουμε την πύλη ώστε οι δήμοι, οι δημόσιες αρχές να καθορίσουν τις προϋποθέσεις ε, στα μέτρα αυτής της επιχείρησης στην οποία θέλουν να θέσουν τελικά τη σύμβαση. Ε, θα καταλήξουμε σε ε, ακριβό σε ακριβή και πολύπλοκη διαδικασία. Αυτό δεν το θέλει κανένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταία σκιώδηση, η κυρία Φόρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολλοί από εμά μιλήσαμε για την πτυχή τη ενέργεια για τι δημόσιε συμβάσει. Θα ήθελα να μιλήσω για τι άλλε αρμοδιότητε τη Επιτροπή, ειδικότερα για την έρευνα και την καινοτομία, Διότι πιστεύω ότι οι δημόσιε συμβάσει αποτελούν κλειδί για την καινοτομία. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα μπορούμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Ε, αυτό θα γίνει, πιστεύω, εν μέρει μέσω τη απλούστευση ε, που θα πρέπει να εξισορροπηθεί όπω το καταλαβαίνω με τη διαφάνεια αλλά και επιτρέποντα επίση, δίνοντα τη δυνατότητα στου ε, αναδόχου όταν παρουσιάζουν μια σύμβαση ή η διατύπωση να αναφέρει ότι προσπαθεί να βρει λύσει για το πρόβλημα αντί να λέει, να καθορίζει ποια θα είναι η λύση, έτσι να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ο ανάδοχος δηλαδή να μην λέει ότι αυτή τη λύση αναζητώ αλλά να λέει αυτό είναι το πρόβλημα και ενθαρρυνώ καινοτόμε λύσει. Πιστεύω ότι οι υποχρεωτικοί στόχοι καινοτομία τη δημόσια συμβάση δεν θα λειτουργήσουν. Δεν γίνεται κατά παραγγελία όλο αυτό. Πιστεύω ότι το να... η απλούστευση θα μας βοηθήσει και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις τοπικές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις επειδή οι μικρότερες επιχειρήσεις θέλουν να προσφέρουν προτάσεις για τοπικές συμβάσεις και όχι διασυνοριακές όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση περάσαμε πολλές ώρες συζητώντα το η χαμηλότερη τιμή δεν είναι η πανάκια ούτε το αναγκάζουμε τις αρχές να αγοράζουν προϊόντα τα οποία ε, μεμονωμένα μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτικά αλλά συλλογικά όχι πρέπει να εξετάζει κανείς και το κόστος κύκλου ζωής και να γνωρίζει ότι πολλές δημοσίες αρχές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση εξέβρεσης ε, μετρητών. Είναι δύσκολο λοιπόν επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. Αλλά ο τομέας κλειδί για τον οποίο θα ήθελα να βοηθήσω είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας, αν μου επιτρέπετε, στις δημόσιες συμβάσεις. Και πιστεύω ότι η αυτή εδώ η Επιτροπή θα πρέπει να ηγηθεί. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει η κυρία Γκροσέτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ε, ήδη και εγκρίνω τα όσα παρουσίασε ο εισηγητής. Όταν συναντάμε διευθύντε ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όταν τι επισκεπτόμαστε, αυτό που ακούμε συνήθω είναι ότι υπάρχει υπερβολικό άχθο, υπερβολική γραφειοκρατία, διοικητική, διοικητικό φόρτο και αυτό είναι που αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Είναι σημαντικό σε εποχέ όπω η σημερινή, σε εποχέ κρίση, να ξαναμελετήσουμε τις ε, ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις και να λάβουμε υπόψη και τις οικολογικές αγορές, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά θα ήταν αντιπαραγωγικό να φορτώνουμε τις ε, βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις μας με επιπλέον περιορισμούς. Φυσικά λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που έχει οριστεί, αλλά ως αντίβαρο θα πρέπει να αλαφρύνουμε το φορτίο που βαρύνει τις επιχειρήσεις μας. Πιστεύω ότι επίσης είναι σημαντικό να επιμείνουμε ιδιαίτερα στην αρχή της αμοιβαιότητας. Ορισμένοι το έχουν ήδη πει. Θα πρέπει να ευνοήσουμε αυτή την αρχή της αμοιβαιότητας ε, ε, όταν δεν εφαρμόζεται αυτή η αρχή, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας ε, θα πρέπει να προτιμώνται από επιχειρήσεις τρίτων χωρών που είναι λιγότερο αξιόπιστες ε, τόσο ε, και δεν πληρούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τα δικά μας. Ε, έχουμε ανισορροπία στον ανταγωνισμό όπως μας επιβάλλεται από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την παραγωγή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί του αθέμητου ανταγωνισμού. Οι κανονισμοί για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να δώσουν κίνητρα για ευρωπαϊκή παραγωγή. Για να ολοκληρώσω ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όλες τις τροπολογίες ε, που υποβλήθηκαν και που επιτρέπουν να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιτρέπουν την υλοποίηση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών που έχουν προβλεφθεί ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Διότι και αυτό αποτελεί μια τεράστια δυσκολία για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε σας. Επόμενος ομιλητής, ο συνάδελφο Βιντάλ Κουάντρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναμφίβολα το πρώτο που έχω να πω είναι να συγχαρώ τον ε, εισηγητή για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι αφιερωμένο σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση των ηλεκτρονικών μέσων. Εγώ βλέπω και με θετικό μάτι και την ενίσχυση της επιτήρησης και την ανησυχία ε, διατήρηση της επιφύλαξης κατά τη διαπραγμάτευση στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Για παράδειγμα, η εφαρμογή των ίδιων κανονισμών στις συμβάσεις με κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και στις συμβάσεις με περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις. Υπάρχουν χώρες στις οποίες ε, το διοικητικό άκθος για τις περιφερειακές αρχές είναι τεράστιο, όπως στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Αυστρία. Και αυτό είναι ουσιαστικά ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη δική μου χώρα. Το έλλειμμα των αυτόνομων κοινοτήτων, των περιφερειακών αρχών. Συνέπεια πρέπει να αφιερώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα υπόλοιπα υποκρατικά επίπεδα που είναι αρμόδια για τις δημόσιες συμβάσεις εφαρμόζοντας κανονισμούς που να προσφέρουν όλες τις εγγύησεις. Ας περάσουμε τώρα στα περιβαλλοντικά κόστη. Όταν υπολογίζονται τα κόστη κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών ε, που αποτελούν τα αντικείμενο δημοσίων συμβάσεων, όταν υπάρχουν παρόχοι υπηρεσιών τοπικοί αυτοί επηρεάζουν τις ε, εκπομπές ε, ε, ρήπων από τις μεταφορές. Θα μπορούσε να υπάρξει διάκριση όμως υπέρ των τοπικών παρόχων. Αυτό δεν μας φαίνεται σωστό. Μετά υπάρχει ένα άρθρο με μια ρήτρα για τον αποκλεισμό της συμμετοχής ενός φορέα σε μια δημόσια σύμβαση. Ωστόσο η διατύπωση είναι αμφίσιμη λέει στα αγγλικά ότι μια αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση οποιονδήποτε οικονομικό φορέα για τον οποίο μπορεί να αποδείξει με οποιοδήποτε τρόπο η αρχή ότι ο ίδιος ο φορέας είναι υπεύθυνος για ε, σφάλματα ε, επαγγελματικής συμπεριφοράς. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχει αμφισημία. Τι σημαίνει αυτό το misconduct, αυτή η επαγγελματική ε, αρνητική συμπεριφορά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι κανόνες πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι και πολύ ακριβείς. Αυτός, αυτή η επιλογή σύνταξης κατά με δεν είναι σαφής. Δηλαδή μπορεί να ε, ερμηνευτεί αυθαίρετα. Θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε τη διατύπωση. Επίσης ε, ήθελα να επαναλάβω ότι το έργο του συναδέλφου ήταν εξαιρετικό και πιστεύω ότι κινούμαστε στο σωστό δρόμο διότι αυτή η οδηγία μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Βέμπερ. Ναι. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το πρώτο πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι ότι στις ε, στην Ευρώπη οι δημόσιες συμβάσεις είναι οι πιο ανοιχτές του κόσμου, είναι ανοιχτές κατά 85%. Ενώ οι κύριοι ανταγωνιστές μας, και δεν μιλάω μόνο για τις αναδυόμενες χώρες, την Κίνα που πάντα προβάλλουμε, αλλά και προηγμένες χώρες όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείες, έχουν δημοσίες συμβάσεις εξαιρετικά προστατευμένες ή και απολύτως ε, ε, μη προσβάσιμες. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Για πόσο καιρό λοιπόν θα αφήσουμε τις δημόσιες συμβάσεις μας ανοιχτές ε, στην προσφόρα που μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε και όχι μόνο από τις αναδυόμενες χώρες, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε αμοιβαιότητα. Αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν το λέω για να κλείσουμε τις αγορές μας. Στι προσφορές από το εξωτερικό, αλλά στο να απαιτήσουμε το άνοιγμα των δικών του αγορών και συμβάσεων. Ε, στις 30 Μαρτίου ε, ένα νομοθετικό νομοσχέδιο για την αμοιβαιότητα των δημοσίων συμβάσεων υποβλήθηκε από την Κομισιόν και θα έρθει σύμφων, ε, σύντομα στο Κοινοβούλιο. Προβλέπει διάφορα εργαλεία διασφάλισης αυτής της αμοιβαιότητας θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να το υλοποιήσουμε. Σε αυτό το κείμενο που μας παρουσιάστηκε εδώ, το οποίο είναι άριστο και υποστηρίζω τις τροπολογίες που υπέβαλαν πολλοί από τους συναδέλφους ε, πριν από μένα, ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα υπόθηκε ήδη, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτό το νέο κανονισμό η ανάθεση τη σύμβασης βάσει της χαμηλότερης τιμής εξακολουθεί ως κριτήριο να διαδραματίζει υπερβολικά σημαντικό ρόλο. Η υπερβολική χρήση ενός τέτοιου κριτηρίου με το χαμηλότερο κόστος, τη χαμηλότερη τιμή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, το έχουμε πει και το επαναλαμβάνω, ε, την καινοτομία και την αναζήτηση, την επιδίωξη καλύτερης ποιότητας και τις καλύτερες σχέσεις ε, ποιότητας και τιμής. Κατά συνέπεια, αυτό το κριτήριο τη τιμής ε, θα πρέπει να αποτελεί ένα κριτήριο μεταξύ των υπολείπων. Και τα υπόλοιπα κριτήρια θα πρέπει επίση να λαμβάνονται πραγματικά υπόψη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, δεν επιμένω γιατί το είπαν και άλλοι, είναι οι διατάξει που έχουν σχέση με την υπεργολαβία. Πρέπει να ενισχυθούν. Ε, Στι μεγάλε δημόσιε συμβάσει, ε, όπω ε, εκείνο ο αυτοκινητόδρομο στην Πολωνία, τον οποίο ανέλαβε η Κίνα μεταξύ του Λούτ και του Βερολίνου, πέτυχαν πολύ χαμηλές τιμές αλλά στη συνέχεια ε, αντανακλάστηκαν αυτές οι μειώσεις τιμών στους υπεργολάβους στην Πολωνία. Έγινε κομμάτια λοιπόν αυτή η συμφωνία διότι αρνήθηκαν οι Πολωνοί αυτές τις ε, εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που τους επιβάλλονταν. Θα πρέπει λοιπόν να ασχολούμαστε περισσότερο με, αυτή την, με αυτά τα διάφορα επίπεδα που συνεπάγεται η υπεργολαβία όταν εκχωρούμε δημόσιες συμβάσεις και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους κυριότερους υπεργολάβους πρέπει να είναι γνωστές πριν από την ανάθεση της σύμβασης και πρέπει να αναφέρονται οι υποχρεώσεις ε, ε, και οι ευθύνες ε, του μέρους ώστε να υπάρχει σαφής και αποτελεσματική επιτήρηση. Στο τελευταίο σημείο διαπιστώνω ότι καταργεί το άρθρο 27 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 27 της τρέχουσας οδηγίας που σχετίζεται με τις διατάξεις για την προστασία της απασχόλησης, της ε, συνθηκών εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος στο νέο νομοσχέδιο. Υπάρχει μια διάταξη για αυτό το θέμα, αλλά η διατύπωσή της ε, μου φαίνεται αρκετά σαφής. Ή σε κάθε περίπτωση ε, πολύ νερωμένη. Ε, γιατί να μην διατηρήσουμε το κείμενο που ήδη υπάρχει και να το εφαρμόσουμε σε όλους τους υπεργολάβους και σε όλη την αλυσίδα προμηθειών. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Βέμπερ. Επόμενος ομιλητής η κυρία Ματσέη Κουκόβιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το σχέδιο γρομοδότησης, Ήταν ώρα να ανανεώσουμε, να αναβαθμίσουμε αυτή την οδηγία. Οι δημόσιες συμβάσεις σήμερα και αύριο, είναι σήμερα και θα είναι και αύριο, πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας νέων και ταυτόχρονα καινοτομίας, ειδικότερα σε εποχές κρίσης ο χρόνος και τα χρήματα είναι το σημαντικότερο πράγμα για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξαιτία αυτού η απλότητα πρέπει να χαρακτηρίζει τα πάντα. Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να αναζητάμε την απλότητα και την ποιότητα ταυτόχρονα. Διότι για τις δημόσιες συμβάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις ε, το μόνο που είχε σημασία ήταν η τιμή, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι η ποιότητα είναι επίσης μια πολύ σημαντική πτυχή. Το ίδιο και η πτυχή της υγείας. Υγεία όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν ε, ε, τεράστια εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τον κύκλο εργασιών τους. Πολύ συχνά αυτές οι απαιτήσει για το πόσο υψηλός πρέπει να είναι ο κύκλος εργασιών ουσιαστικά αποτελεί κλειστέ πόρτε, κλείνει τι πόρτες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή την ε, βελτίωση της οδηγίας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας με αυτή την νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις ε, που άκουσα από τους διάφορους προλαλήσαντες, ε, από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, επί δύο θεμάτων. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις ΜΜΕ. Θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη πολλέ συζητήσει και πολλά ψηφίσματα μάλιστα που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο. με μια ζήτηση που είχαμε με τον προκάτοχο του Μπισελ Μπαρνιέ, τον κύριο Σελίμ Μπακλεβί, στον οποίο είχαμε ζητήσει με ισχυρή πολιτική πλειοψηφία να επαναδιαπραγματευτεί την συμφωνία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Εθνή Οργανισμό Εμπορίου και νομίζω ότι τότε κάναμε ένα τεράστιο λάθος. Ε, δεχθήκαμε αυτή την εξαίρεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δημόσιας συμβάσεις και εκείνη την εποχή είχαμε ζητήσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δεν ξέρω αν ο σημερινό Επίτροπο Εμπορίου θα το δεχόταν, αλλά προ τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι εδώ την οδηγία. Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να βρούμε μια διατύπωση που να βρίσκει σύμφωνα όλα, σύμφωνα σε όλες τις πολιτικές ομάδες ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και αυτό στο σύνολο των απαιτήσεων διότι αυτό που πρότεινε η Κομισιόν το να περιορίσουμε τον αριθμό της απαιτήσει εγγύησεων, όλα αυτά είναι πολύ καλά, ωστόσο αυτό δεν θα εμποδίσει τις εξελίξεις που διαπιστώνουμε, που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε εξής, οι μεγάλες επιχειρήσεις, ε, ουσιαστικά παίρνουν τα πάντα από όλε τι δημόσιε συμβάσει, ε, ε, παίρνουν υπεργολάβου του οποίου πληρώνουν πολύ άσχημα, αυτές ε, πτωχεύουν και μετά τις ε, ξαναγοράζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και μετά δεν υπάρχει ανταγωνισμός και ανεβαίνουν οι τιμές. Πρέπει λοιπόν να, να παρακολουθούμε τη λειτουργία αυτών των αγορών και να μπορέσουμε να δώσουμε μια σωστή θέση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μιλάω για ποσοστώσεις, γιατί όχι, διότι πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μια διατύπωση ώστε να δώσουμε μια πραγματική θέση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε με ένα κανονισμό για την υπεργολαβία είτε πρέπει να συμφωνήσουμε για τροπολογίες οι οποίες επιβάλλονται στα κράτη-μέλη. Δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά την αμοιβαιότητα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιτύχουμε πολιτικές πλειοψηφίες ε, για την απέτηση αμοιβαιότητας. Αγνοούσα και ευχαριστώ τον συναδελφό Βέμπερ που μας ενημέρωσε ότι υπήρχε μια άλλη νομοθετική διαδικασία δεν ξέρω πώ όλα αυτά θα συντονιστούν, αλλά αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να συμφωνήσουμε για μία διατύπωση μιας συμβαστική τροπολογίας. Νομίζω στο ε, άρθρο 55 θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εντολοδόχος θα μπορεί να αποκλείσει ένα συμμετέχοντα ή μία επιχείρηση στη χώρα καταγωγή, ε, της οποίας χώρα καταγωγής δεν έχει κανόνες παρόμοιους ανοίγματο των δημοσίων συμβάσεων ενδεχομένω με τριμερή διάλογο, χρειαζόμαστε συνοχή, αλλά για να έχουμε πολιτική πλειοψηφία πρέπει να τονίσουμε ότι απαιτούμε αυτή την αμοιβαιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει τον ε, ανταγωνισμό ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι δημόσιες συμβάσεις και γι' αυτό είναι αποφασιστικής ε, σημασίας. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκιουρκ και τον ευχαριστώ για την λεπτομερή του ανάλυση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε πώς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου δημιουργούνται και οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης, διότι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια το 80% των ε, θέσεων απασχόλησης ε, ε, δημιουργείται σε τέτοιες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς τους μεγάλους διαγωνισμούς μπορούμε να τους χωρίσουμε σε μικρότερα κομμάτια. Πιστεύω ότι οι δημόσιες αρχές ε, θα πρέπει να ε, εκπονούν ε, πιο αναλυτικά τις, τους διαγωνισμούς. δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσουμε αυτό στο τελικό κείμενο, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια προσέγγιση. Όχι να δώσουμε ποσόστοση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς, αλλά να τις ενθαρρύνουμε χωρίζοντας τις μεγάλες συμβάσεις σε μικρότερα κομμάτια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουν τελειώσει οι εγγεγραμμένοι για να μιλήσουν. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Κρακούν. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Εγώ έχω μόνο δύο-τρεις παρατηρήσεις να προσθέσω σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε σήμερα για την έκθεσή σας. Πρόκειται για το πιο πολυσυζητημένο θέμα. Οι δημόσιες συμβάσεις. Επομένως, στο νομοθέτημά μας θέλω υπόψη αυτά τα οποία είπατε. Κάθε φορά κανείς καταλήγει στο ότι με την οδηγία θα πρέπει να έχουμε ένα νομοθέτημα που να μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε διαφάνεια. Να έχουμε επομένω ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε οι αρχές να μπορούν να εξετάσουν κάθε φορά την πράσινη πλευρά της ε, σύμβασης. Δεν πρέπει να καθίσουμε από τώρα στο τι θα αγοράζει κάθε φορά η κρατική αρχή. Α είμαστε ρεαλιστέ, μπορούμε πούμε θα αγοράζετε μόνο πράσινα ή 20% πράσινα ή κάτι άλλο τέτοιο. Άρα θέλουμε να δίνουμε μια νομική βάση και μετά να συνδέουμε την νομική βάση με τις διάφορες ε, πολιτικές και τις διάφορες οδηγίες που υπάρχουν. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει οδηγία για το περιβάλλον κλπ. Οπότε θα πρέπει να αναφέρεται κανείς σε κάθε σύμβαση ε, σε αυτά τα νομοθετήματα, να παραπέμπει τον, η σύμβαση κρατική εκεί πέρα. Και οπότε ε, να ακολουθούν την πολιτική μας οι διεξάγοντες του διαγωνισμού, οι αρχές. Δεν μπορούμε εμείς να τους πούμε από τώρα τι θα κάνουν. Επομένως, έχουμε τις πράσινες ε, κρατικές συμβάσεις για τις οποίες σκεφτήκαμε ότι ε, με την εξέλιξη των πραγμάτων ότι οι αρχές συχνά θεωρούν ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα να αγοράσουν πράσινο προϊόν ή δεν ξέρουν τι γίνεται. Γι' αυτό και εμείς ε, εδώ βάλαμε μία διάταξη ούτως ώστε με κάποια κέντρα ενημέρωσης να βοηθούνται να επιλέξουν τα πράσινα προϊόντα ή τις πράσινες υπηρεσίες οι αρχές. Γι' αυτό και η σημασία η τροπολογία που λέει ότι οι αρχές θα πρέπει να στρέφονται προς αυτά τα προϊόντα, αλλά πάντως είναι δύσκολο να το επιβάλλουμε. Λοιπόν, θα υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες εθνικές που έχουν το ρόλο αυτό. Για τη διαπραγμάτευση τώρα δούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα να υπάρχουν πρώτες και περισσότερες ίσως να μην υπάρχουν δεσμενείς διακρίσεις να υπάρχει ε, διαφάνεια θέλουμε και είναι δύσκολο να έχουμε ανοιχτή διαπραγματεύση σε κάθε περίπτωση γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε κατάχρηση Άρα, να έχουμε περισσότερες διαπραγματεύσεις από ότι προέβλεπαν οι οδηγίες του 2004 αλλά οι διαμετρήσεις αυτές να ε, γίνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επίσης τώρα, όσο αφορά την αμοιβιότητα όπως αναβάλλατε, υπάρχει συγκεκριμένο νομοθέτημα το οποίο πρόσφατα προτάθηκε και στα πλαίσια εκείνου του νομοθετήματος θα το συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν εδώ εμπλεκόμενα, αντιμαχόμενα συμφέροντα. και τέλος πάντων το συζητούμενο σήμερα νομοθέτημα δεν είναι η κατάλληλη ώρα να την αμοιβαιότητα, πάντως είναι κάτι σημαντικό και θα το δούμε. Ωραία, λοιπόν, το συμπέρασμα αυτής της συζήτησης που ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θέλατε το λόγο? Ε, Ευχαριστώ. Μήπως ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορούσε να εξηγήσει αυτό το τελευταίο που είπε, γιατί τώρα να μην ε, συζητήσουμε, να μην ε, ρυθμίσουμε κάτι για την αμοιβαιότητα. Ναι, θέλετε, σας παρακαλώ να ξαναπάρτε το λόγο και να απαντήσετε σε αυτό την ερώτηση, να εμβαθύνετε λίγο. Ναι, φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στι διαπραγματεύσει του Διεθνού Οργανισμού Εμπορίου. Για αυτόν τον τομέα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία. Έχουν ξεκινήσει εδώ και, καιρό, και καιρό οι διαπραγματεύσεις. Ε, βρίσκονται εν εξελίξη και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τεχνικά έτοιμοι να το πράξουμε αυτό σε αυτή την πρόταση το λόγο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί ξεχωριστό ε, νομοθέτημα για το θέμα αυτό. Διαφορετικό από τις οδηγίες. Ε, μισό το περίμενα για να ακούσω το τέλος της διερμηνίας. Κύριε Οντή, για το λόγο. Πρόεδρε, ο κύριος Οντή. Ε, ε, είμαστε ανοιχτοί από παντού. Και όλοι θα σας πούνε, δεξί, αριστερή, πολιτική, μην είσαστε αφελείς. Μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ. Και πόσο καιρό θα κάτσει αυτό, έναν αιώνα. Και τι θα γίνει. Όταν τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις θα έχουν πεθάνει οι ΜΜΕ και η, και η βιομηχανία. Επομένως, τι γίνεται. Θα πρέπει να, να είμαστε συμβατοί με τον ΠΟΕ. Ε, γιατί ε, θεσπίζεται κάποιου κανόνες, ε, προσφεύγουμε τα στον ΠΟΕ οι εταιρείε και πάει. Τι θα κάνουμε. Ε, φταίμε εμεί, αλλά φταίτε και εσεί. Εμεί σα τα λέμε, δεν μα ακούτε. Ε, αυτή η απάντηση δεν είναι απάντηση που είπατε. Εμεί ε, ελπίζω ότι θα έχουμε την ε, κατάλληλη πλειοψηφία, ούτω ώστε να γίνει κάτι όπω είπε ο κ. Βέμπερ και για την ε, Δεν θέλουμε να είμαστε αφελεί. Ακούστε επιτέλου και του πολίτε. Ο συνάδελφος Βέμπερ, έχετε το λόγο, ναι. Ε, μια πληροφορία, διότι παρακολούθησα αυτό το ζήτημα αυτό που προτείνεται, αυτό που συζητιέται σε αυτό το νομοσχέδιο για την αμοιβαιότητα Μιλάμε για, συζητιούνται τρία μέσα, τρία εργαλεία τα οποία δεν υπάρχουν και ακόμα πρέπει να επιτύχουμε την πλειοψηφία για να τα επιβάλλουμε. Ε, κατά με είμαστε μακριά. Το πρώτο εργαλείο επιτρέπει τοπικούς ε, υπευθύνους ε, ανάθεσης συμβάσεων, δηλαδή εντολοδόχους οι οποίοι μπορούν να μην ανοίξουν τι δημόσιες συμβάσεις τους σε χώρες με τις οποίες δεν υπάρχει αμφιβεβαιότητα. Αυτό είναι το πρώτο εργαλείο. Το δεύτερο εργαλείο είναι η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κλείσει τις δημόσιες συμβάσεις για τις χώρες που κλείνουν τις δικές τους προς Και το τρίτο εργαλείο και αυτό το γνωρίζετε ήδη διότι ήδη ε, εφαρμόζεται να κλείσουμε την πρόσβαση στις αγορές μας σε υπερβολικά παράλογα χαμηλές προσφορές. Το φίλτρο αυτό το ασκούν οι τοπικές αρχές. Αυτά έχουμε στο τραπέζι. Δεν έχει ψηφιστεί. Εκεί που συμφωνώ με τους, φίλους, με τους συναδέλφους μου είναι ότι σίγουρα έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο συζητιέται και ελπίζουμε ότι όλο αυτό θα ψηφιστεί και θα ενισχυθεί, αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει στο κείμενο ε, στο οποίο ψηφίζουμε εμείς να, δεν, μας, δεν μας εμποδίζει να τα εντάξουμε ήδη αυτά τα εργαλεία. Ναι, κύριε Λάγκεν. Μία σύντομη ιστορία από την ιστορία των δημοσίων συμβέσεων να σας πω. Ε, το 1996 ήμουνα νέος ε, ευρωβουλευτής και συμμετείχα σε διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις ε, και το πρώτο νομοσχέδιο του Μόντι την πρόταση αυτήν την υιοθέτησε το Κοινοβούλιο με 400 απέρριψε μάλλον την πρόταση με 430 ψήφους κατά δύο και γιατί λόγω της έλλειψης αμοιβαιότητας. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Ως Ιταλίδα πολίτης ε, θα ήθελα να μην το διηγήσετε και πολύ έξω αυτό το επεισόδιο, εντάξει. Λοιπόν, τα τελικά συμπεράσματα στον συνάδελφο Γκίρκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τους συναδέλφους ε, για αυτή την ε, πολύ πλούσια συζήτηση που εμπλουτίζει την αμοιβότητα με νέα στοιχεία. Και χωρίς όμως αυτά η συζήτηση θα ήταν άριστη και θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για το ε, μελλοντικό μας έργο. Φοβάμαι ότι Υπάρχουν πολλές, πολλές τροπολογίες, αλλά αν ακολουθούν την κατεύθυνση την οποία διακρίνω εγώ, θα βελτιώσουν πράγματι το τελικό κείμενο. Δεν θέλω ακόμα να απαντήσω λεπτομερώς ε, ε, σε κάθε τροπολογία ε, και σε κάθε σχόλιο. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για τη συμβολή του. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία πράγματα και να απαντήσω σε αυτά. Πρώτον, η εμφάνιση της κοινωνικής πτυχής στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων όπως προτείνεται από το συναδέλφο μου Μπαλσίτης. Δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο διότι χρειάζεται ε, ισορροπία, εξισορρόψη με την οικονομική αποδοτικότητα. Περιμένω τροπολογία αλλά αμφιβάλλω όπως και ο συνάδελφος Λορά, ε, δεν ξέρω αν οι δημόσιες συμβάσεις είναι ο καλύτερος τομέας για να αναδείξουμε την κοινωνική πτυχή. Δεύτερον, η ενεργειακή απόδοση, ε, η εμφάνιση δηλαδή της άποψης των πρασίνων, της πράσινης άποψης. Εγώ το έχω θέσει αυτό στο επίκεντρο της γνωμοδότησής μου. Χαίρομαι που η κυρία Αλσή ε, αντέδρασε. Είπε ότι η εκθέση θα πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά αυτό το σημείο εγώ θεωρούσα ότι ο συμβιβασμός που είχε επιτευχθεί μέσα σε άκρες όσον αφορά την, οικονομία, ε, την ενεργειακή απόδοση, εγώ πήρα αυτή, αυτό το συμβιβασμό και τον ενέταξα στην γνωμοδότησή μου. Είναι το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω και θα χαρώ να δω οποιαδήποτε πιθανή τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω ένα σημαντικό σημείο της συζήτησης ε, πριν από λίγο. Συμφωνώ ότι η ίση μεταχείριση πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο. Προς το παρόν δεν υπάρχει. Αν έχετε τροπολογίες θα είναι ευπρόσδεκτες. Θεωρώ ότι όσα μας είπε η Κομισιόν θα πρέπει να μας οθήσουν να αναπτύξουμε αυτή την ιδέα και να την εντάξουμε στο τελικό κείμενο. Αναμένω λοιπόν τις τροπολογίες της κ. Κλωσάρ, του κ. Ντί. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλες τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ όλους που συζητήσαμε όλοι μαζί και έχουμε το χρόνο μέχρι την Δετάρτη για να υποβάλουμε τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ωραία, λοιπόν, Να κλείσουμε και αυτό το σημείο τη ημερήσιας διάταξη. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που μίλησαν για την ποιότητα αυτή τη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 6 Ιουνίου, 12 η ώρα το μεσημέρι επόμενο σημείο. Ε, ελπίζω γι' αυτό να τηρήσουμε καλύτερα τους χρόνους. Αφορά τι συμβάση που συνάπτει από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η συγητή, ο συνάδελφο Μπαλτσίτη, τον οποίο δίνει αμέσω το λόγο για την παρουσίασή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Μόλις ολοκληρώσαμε την ε, συζήτησή μας για τις αρχές ε, που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Εγώ είμαι συντάκτης γνωμοδότησης σχετικά με την ε, οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ίδατος της ενέργειας των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Υπάρχουν δύο οδηγίες που διέπουν τις δραστηριότητες αυτούς τους τομείς. και θα ήθελα να τονίσω ότι οι περισσότερες συμβάσεις... Θα ήθελα να, να, να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικός ο όγκος των συμβάσεων στους τομείς αυτούς. Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλή η πρόταση της Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ιδιομορφίες του τομέα αυτού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το επίπεδο απελευθέρωσης ε, στους τομείς αυτούς ε, διαφέρει από κράτος μέρος σε κράτος μέλος. Η Κομισιόν είχε δημόσιες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους. Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφωνούν ομόφωνα ότι οι, κανόνες, οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν για ε, τους τομείς κοινή ωφελίας θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και να, διότι αντικατοπτρίζουν τις ιδιομορφίες αυτών των τομέων. Ε, υπάρχει ακόμα μεγάλη συγκέντρωση και υπάρχει έλλειψη ε, ανταγωνισμού στον τομέα αυτών για ιστορικούς, ε, αυτό οφείλεται σε ιστορικούς λόγους μπορεί να ε, αποδοθεί και σε γεωγραφικούς και άλλους λόγους Γι' αυτό η Επιτροπή έχει υποβάλει την πρόταση αυτή. Ε, ωστόσο, με τις αλλαγές που βλέπουμε, με το άνοιγμα των αγορών, θα αλλάξουν και οι κανόνες που διέπουν ε, τους τομείς αυτούς. Θα ήθελα τώρα να φτάσω στην ουσία της πρότασης της Κομισιόν. Καταρχήν, η πρόταση αυτή ε, εισάγει τροποποιημένους ορισμούς των ε, βασικών ενιών λαμβάνοντας υπόψη την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπως ε, είναι η φορείς δημοσίου δικαίου, καθώς και η έννοια ε, των δημοσίων ε, συμβάσεων. Ε, η πρόταση επίσης κάνει διάκριση ανάμεσα σε υπηρεσίες προτεραιότητας και μη προτεραιότητας. Θέλει να επιλέξει καινοτόμε διαδικασίες και θα πρέπει αυτοί που υποβάλλουν προσφορές να μπορούν να επιλέξουν από έξι λύσεις ένα από τα σημαντικότερα επιτέγματα μας κατά τον εξυγχρονισμό ε, του τομέα των δημοσίων συμβάσεων είναι οι ηλεκτρονικές συμβάσεις. Όταν εισαχθούν οι ηλεκτρονικές ε, δημόσιες συμβάσεις θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους ε, θα απλοποιήσουμε τη διαδικασία και αυτό θα ε, είναι προς, ε, προς μεγάλο όφελος ε, των μεσαίων επιχειρήσεων που θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων. Προβλέπεται υποχρεωτικό σύστημα υποβολής κοινοποιήσεων σε ηλεκτρονική μορφή και επίσης υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των, διανομή των εγγράφων του διαγωνισμού. Θα ήθελα να προτείνω να αλλάξουμε τις ε, προθεσμίες που προτείνει η Κομισιόν, διότι είναι υπερβολικά σύντομες. Οι φορείς που συμμετέχουν ε, στους δημοσίους διαγωνισμούς θα πρέπει να ε, προσαρμοστούν. Η πρόταση μιλάει και για τις κοινωνικές στοιχές των δημοσίων συμβάσεων αναφέρεται η δυνατότητα απαγόρευσης ε, ε, συμμετοχής ε, σε κάποιους φορείς εάν σημειώνονται παραβιάσεις. Επίσης θα πρέπει να επιτρέψουμε τη διεξαγωγή καινοτόμων δημοσίων συμβάσεων και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την τυχή που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Η δυνατότητα αυτή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα ε, υπάρξει όμως μόνο όταν ε, όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόσουν την ηλεκτρονική διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι οι κανόνες που ισχύουν στα κράτη-μέλη διαφέρουν. Στην πρακτική εφαρμογή ε, θα ε, είναι πιο καθαρά τα προβλήματα. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ομοιομορφία σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να ξεκινήσουμε από τους αισιόδης εισηγητές, ο κύριος Λάνιεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος εδώ. Έχουμε την συνέχιση ε, κανόνων δημοσίων συμβάσεων που έχουν αποδείξει την αξία τους. Ε, ένα πρόβλημα που συζητιέται ακόμα είναι πώς μπορούν να συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο συντάκτης της νομοδότησης έχει υποβάλει ε, προτάσεις, θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις αυτές. Όσον αφορά την παράταση των προθεσμιών, δεν είμαι βέβαιος μήπως τελικά είναι πολύ μακρά η διαδικασία διότι προτείνεται σημαντική παράταση των προθεσμιών. Θα πρέπει να συζητήσουμε μήπως η πρόταση της Κομισιόν είναι τελικά σωστή. Δύο πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Καταρχήν, ε, τα κατόφλια που δεν έχουν αλλάξει εδώ και 20 χρόνια παρά την εισαγωγή του ευρώ και ε, επίσης το 3% των ε, συμβάσεων ε, ανατίθενται διασυνοριακά στην Ευρώπη. Ε, υπάρχουν δηλαδή κανόνες για την διεξαγωγή των διαγωνισμών σε διασυνορικό επίπεδο, αλλά οι επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από αυτό σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην πρόθεσή μας να συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματικότητα. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον μηχανισμό. Μήπως μπορέσουμε με κάποιο νέο τρόπο να αλλάξουμε το μηχανισμό αυτό. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, η Κομισιόν ε, έχει ε, εισάγει ε, υποχρέωση κοινοποίησης ε, και κατόφλια και θα πρέπει να εξετάσουμε αν αυτό αιτιολογείται. Και έχω ερωτήσεις σχετικά με τον κύκλο ζωής, ε, μήπως ε, θα πρέπει να το ε, συμπεριλάβουμε αυτό και ο συνάδελφος Ταραμπέλα στην ΙΜΚΟ πρότεινε να συμπεριλάβουμε ένα σωρό ιδέες από τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων όχι μόνο κανόνες δηλαδή, ε, αλλά μπορούμε ε, έτσι να, στους υποβάλλοντες προσφορές ε, να επιβάλλουμε υπερβολικό άχθος. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα οι αρχές που διεξάγουν τους διαγωνισμούς να είναι υποχρεωμένες να εξετάσουν και εναλλακτικέ ε, προ, ε, προτάσεις, προσφορές. Ε, η Κομισιόν λέει ότι μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά εγώ λέω ότι θα πρέπει να το κάνουν αυτό και το θέμα της ε, φτηνής τιμής ε, δεν είναι ο μόνος ε, παράγοντας. Μπορεί να υπάρχουν τεχνικά πιο πολύπλοκες λύσεις οι οποίες θα πρέπει να εξετάζονται. Επίσης, στην οδηγία αυτή πιστεύω ότι κάπου θα πρέπει να έχουμε την υποχρέωση για τα κράτη-μέλη, για διαγωνισμούς σε κάτω από το κατόφλι, ε, να είναι υποχρεωμένα να ε, λαμβάνουν υπόψη τις ε, ίσες συνθήκες ανταγωνισμού, την μη διάκριση και την πρόσβαση σε όλους θα πρέπει σε κάποιο άρθρο υπό κάποια μορφή να συμπεριλαμβάνονται αυτά. Ε, οι ευρωπαϊκοί κανόνες υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο. Πολύ όμως και στην Γερμανία, όπου λόγω της ομοσπονδιακής δομής είναι ακόμα πιο δύσκολο, Ε, ε, θεωρείται ότι από ένα συγκεκριμένο κατόφλι μόνο ισχύουν οι ε, ευρωπαϊκοί κανόνες. μου φαίνεται ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις βασικές αρχές του πρωτογενούς δικαίου και εδώ. να θυμόμαστε ότι πρόκειται για γνωμοδότηση, όχι για οριστική έκθεση, αλλά θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τη θέση μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Φιώνα Χόλ. Ευχαριστώ πολύ. Εισήγητα για την εκθεσή σας. Επιτρέψτε μου όμως κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα πρώτα, αυτό το, το κόστος το συνδυόμενο με τον κύκλο ζωής. Είναι από τα πιο αποτελεσματικά πράγματα που έχουμε στη διαθεσή μας ε, αυτές οι συμβάσεις τόσο ώστε να μπορέσουμε να οθήσουμε του ε, τους ε, στόχους που θέλουμε την βιομηχανία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να δούμε ε, τι έχει προβλεφθεί στο παρελθόν σχέση με σήμερα, σε σχέση με αυτές τις συμβάσεις, γιατί τελικά δεν θέλουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε την ενεργειακή οδηγία, διότι το, το, ο βαθμός της συμμετοχής δεν είναι ο ίδιος. Η ενεργειακή οδηγία ασχολείται με τις λεπτομέρειες. Τώρα όμως έχουμε μια, μια γενικότερη αντιμετώπιση, άρα και το ένα και το άλλο είναι χρήσιμα και ρυθμίσεις και στη μία στην άλλη οδηγία. Επίσης, ε, συμφωνώ ότι οθεί προ και προς καινοτομία η δημοσία σύμφωνη ιδίω, εάν είναι προσεγμένες οι συμβάσεις και αν έχουμε μια ε, ανοιχτή προσέγγιση προς την ε, καινοτομία. Τώρα είναι θέμα των κρατών μελών. Και θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ρύθμιση πάντως. Όσον αφορά το, το κόστος, η ρύθμιση για το κόστος ε, του κύκλου ζωής. Και τελικά οφειλημένο δεν είναι μόνο το περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη. Αυτό το τονίζουν διάφορες μελέτες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση μέχρι και 20 δις ευρώ ετησίως. Δεύτερον, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές, τα ηλεκτρονικά μέσα, ναι, είναι πάρα πολύ θετικό έτσι απλουστεύεται το σύστημα, έτσι περιορίζεται το κόστος. Σύμφωνο με αυτά που είπε ο συγητής. Τα κρατημέλη πρέπει να εφαρμόσουν τον κώδικα των ίστων πρακτικών και να διευκολύνουν την προσβασιμότητα στις ε, συμβάσεις μία ΜΜΕ και τα κρατημέλη θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον κώδικα διοντολογίας. Αξίζει να δίνουμε την ευκαιρία στις ΜΜΕ να μάθουν γιατί δεν εφαρμόζεται ο κώδικας. Τέλος. Κάτι το οποίο ε, λέει εδώ η Κομισιόν που λέει για κάποια εποπτική εθνική αρχή που θα κατευθύνει κλπ. Αυτό είναι προβληματικό. Πρέπει να γνωρίζουμε τι κάνουν άλλες χώρες θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει ε, διάχυση των πληροφοριών, αλλά δεν θέλουμε σε καιρό κρίσης να έχουμε ακόμα μια υπηρεσία που θα αναλώνει χρήμα. Μήπως μπορεί να γίνει οικονομικότερα ε, το ίδιο. Ίσως ε, οι εθνικές αρχές να το κάνουν αυτό. Όπως γίνεται και σε άλλους τομείς, ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες. Αντί δηλαδή να συγκροτείται μια νέα υπηρεσία, να έχουμε τις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές που να αναλαμβάνουν αυτό το έργο της εποπτείας. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για την αξιόλογη εκθεσή του. Δεν ζητήσει άλλο το λόγο. Τώρα θα τον δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις, για τα σχόλια. Θα ληφθούν όλα υπόψη. Πάντως έχω δύο-τρεις παρατηρησούλες σε σχέση με αυτά που άκουσα. Βεβαίως και ήδη έχουμε κάποιες διατάξεις για τις ΜΜΕ, για τις βοηθήσουμε σχέση με τις συμβάσεις και θα συνεχίσουμε την βελτίωση του κειμένου. Πάντως, θέλω να πω κάτι για τις διασυνοριακές τέτοιες συμβάσεις. Ότι πάντοτε μας γνωστοποιείται ότι μόνο το 3% γίνεται στην εσωτερική αγορά Δηλαδή, ε, λίγα πράγματα. Έτσι λένε οι στατιστικές μας διάθεσή μας όσον αφορά επομένω ε, τις άμεσες διασυνοριακές συμβάσεις. Να γίνεται στο ένα κράτος μέλος η σύμβαση και να εκτελείται αλλού. Έχουμε δηλαδή κάποιες εταιρείε που συνεργάζονται με κάποια άλλη που βρίσκεται αλλού ή έχει κάποια θηγατρική και αυτό φτάνει το 13% των συμβάσεων που γίνονται πάντως από ό,τι γνωρίζουμε στην ιστορική αγορά υπάρχει μπορεί να γίνει μεγαλύτερη συμμετοχή και γι' αυτό και έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις. Πώς θα υπάρχει μια ξεκάθαρη ρύθμιση για να οργανωθεί καλύτερα αυτή η, η μορφή συμβάσεων, ιδίες συνοριακές. Επίσης, προτάθηκαν ε, προθεσμίες ελαστικότερες, πιο μεγάλες από όσο προτείναμε εμείς. Έχουμε τάξει αυτές τις προθεσμίες για να υπάρχει αρκετή διαφάνεια για να υπάρχει... Μην, μην, μην αποκλείσουμε τις θεσμενείς διακρίσεις. Μπορούν οι αρχές να τάξουν προθεσμίες μεγαλύτερες. Εμείς είπαμε ποιο είναι το μήνυμο. Αυτά και σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Βαλτσίδης μπορείτε να κλείσετε σε σχέση με την αξιόλογη έκθεσή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους για τις χρήσιμες συμβουλές τους. Όσον αφορά τις προθεσμίες, δεν νομίζω ότι είναι ουσιαστικό στοιχείο της πρότασης. Έχει γίνει συντονισμός με, τη βασική, με την ε, αρμόδια της Ουσίας Επιτροπή και συζητάμε το θέμα αυτό με αυτήν. Είναι σημαντικό το ότι μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικές εμπειρίες ε, τους ε, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Εγώ συμμετείχα στη διαμόρφωση του τομέα αυτού στην χώρα μου και καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό εφαρμόσαμε κάποιες ε, εξαιρέσεις. Αυτό είναι φυσικό ε, σε μια τέτοιου τύπου διαδικασία. Ε, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν συμφωνούν με κάποια στοιχεία, με κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω την Επιτροπή, ιδιαίτερα το, το τμήμα που έχει να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις, να να προσπαθήσει να συγκεντρώσει τις εμπειρίες διαφορών κρατών μελών. Ε, αναφέρθηκα στην ε, οδηγία περί υπηρεσιών και ε, στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας οι διάφορες χώρες ε, εφαρμόζουν διάφορες πρακτικές. Θα πρέπει, πιστεύω, να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας ε, και σιγά-σιγά θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω όλους μας να υπερασπιστούμε την αγορά μας, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, να χάσουμε θέσεις απασχόλησης, να χάσουμε ε, δημόσια έσοδα, φορολογικά έσοδα, διότι οι προκλήσεις στον τομέα του ανταγωνισμού είναι σημαντικές. Ε, αντιμετωπίζουμε ανταγωνισμό από χώρες που δεν εφαρμόζουν τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είπαμε ότι έχουμε αυτή την, ε, την προθεσμία στις 6 Ιουνίου του το μεσημέρι και όπως και στο παρελθόν είπαμε θα ολοκληρώσουμε λίγο πιο νωρίς Έχουμε ένα τεταρτάκι που τελειώσαμε πιο νωρίς και θα συνεχίσουμε ξανά στις 3.